Καλημέρα. Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη καταρχάς. Σημείο 31. Ψηφίζουμε την έκθεση Γκαμπριέλ. Μάλλον αυτό είναι το σημείο. Έφτασε επιστολή από την Κορεπέρα εν τω μεταξύ. και ίσως διεξαχθεί αυτή η ψηφοφορία που ε, αναφέρεται ως πιθανή 35 το σημείο 35 αναβλήθηκε 36 σχέδιο γνωμοδότηση για τι διαπραγματεύσει για του σχετικού φακέλου με το ποτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τα μαθήματα που μπορούμε να συναγάγουμε προσετέθη στην ημερήσια διάταξη. Και νέο σημείο έχει προσθεθεί για τις 13 Φεβρουαρίου, δηλαδή αύριο, 9 με 10 η παρουσίαση της εκθέσεως ε, Κοέλιο για την, ε, τον έλεγχο των εξωτερικών συνόδων και σημείο 36 Αργεντίνη. Ε, λοιπόν, η καταπολέμηση της, του ξεπλήματος χρήματος θα αναβληθεί για τις 20 Φεβρουαρίου. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, Λοιπόν, έχουμε τις συστάσεις των συντονιστών. Συντάχτες Κίνγκεγκάρτς, έκθεση για την Επιτροπή Προπολογισμών και τι διαπραγματεύσει του ποτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αντιρρήσει δεκτών. Γλωσσική κάλυψη. Δεν έχουμε φιναδικά, εσθονικά, μαλτέζικα και κροατικά. Σήμερα δεν έχουμε διερμηνία από αυτές τις γλώσσε. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Εγκρίνουμε τα πρακτικά του 27 και 28 Νοεμβρίου. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Πάμε στο σημείο 4. Έγκριση διορθωτικού για, την ανταλλαγή, για πρόγραμμα ανταλλαγής και βοήθειας που παρέχεται για την, της κυρίας Μακεντάρη που αφορά την καταπολέμηση παραχάραξης του ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 216 του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου, και μετά από τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υθετήθηκε στην πρώτη ανάγνωση τον περασμένο Δεκέμβριο, ο κανονισμός που αποφασίζει την ανταλλαγή, κατάρτιση ε, και το σχετικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση παραχάραξης του ευρώ θα διορθωθεί η απόφαση μέσω διορθωτικού κειμένου. Συμφωνείτε, η είναι η κυρία Μάκινταρ. Έχετε να πείτε κάτι κυρία Μάκινταρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σωστά τα είπατε. Ψηφίσαμε και πιέσαμε να εξεταστεί από την Ολομέλεια το ταχύτερο δυνατόν. Μας είπαν ότι αν πιέζαμε να μπει στην ημερήσια διάταξη, έπρεπε μετά να περάσουμε το διορθωτικό, δεν άλλαξε τίποτα. Οι γλωσσομαθείς νομικοί άφησαν το κείμενο είχε. Είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Ήδη ψηφίσαμε την πρόταση, ψηφίσαμε στην Ολομέλεια. Απλώς πρέπει να κάνουμε την τυπική διαδικασία και να το εγκρίνουμε, το διορθωτικό κείμενο. Ευχαριστώ κυρία Μάκιντάρ. Εντάξει, έτσι. Τελειώσαμε αυτό και μπορούμε να πάμε στο σημείο 5. Αφορά την όλη κατάσταση των διοργανικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο νομοθετικών διαδικασιών. Η κυρία Μακιντάρ είναι η συγγήτρια και όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. για την οδηγία για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων κατά της παραχάραξης ε, μέσω ποινικού δικαίου να εφαρμοστεί αυτή η προστασία. Η κυρία Μάκιντάιρ μας ενημερώσει. Ευχαριστώ λέει, κυρία Μάκιντάιρ. Είμαι ευγνώμων προς όλους τους κοιόδης για τη βοήθειά τους και τη συνεργασία τους. Είμαστε το μέσο τριμερών διαλόγων. Προχωράμε αρκετά καλά. βρήκαμε κοινό έδαφος στα περισσότερα ζητήματα και έχουμε και άλλο τριμερή διάλογο σήμερα το βράδυ. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθούν όλα τα ζητήματα σε αυτή τη φάση. Ελπίζω, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Ίσως χρειαστούμε και περιττέρω προσπάθειες. Μετά από αυτό όμως φαντάζομαι μέσω γραπτής διαδικασίας μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία. Τι να πω. Πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Ελληνική Προεδρία και ελπίζω να διεκπαιρωθεί το όλο θέμα τάχιστα. Ευχαριστώ κυρία Μακιντάρ για αυτή την παρουσίαση. Τελειώσαμε και με αυτό. Οπότε μπορούμε να πάμε στο σημείο 6, ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Ευρωπαϊκή Ένωση Λίζα, κύριο Κρουμ Γκάρκοφ. Εκτελεστικός διευθυντή του οργανισμού που είναι υπεύθυνο για υπηρεσιακή διαχείριση μεγάλη κλίμακα συστημάτων πληροφορική το σύστημα πληροφορικής, το SAS2 του Σέγγεν, το σύστημα ενημέρωση για για τη θεώρηση και το Eurodac. Ας μας ενημερώσει λοιπόν ο κύριος Γκάρκοφ για τα βασικά επιτεύγματα του περσινού έτους και τις προβλεπόμενες εξελίξεις για τον επόμενο χρόνο. Και έχετε το λόγο κύριε Γκάρκοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να έλθω ενώπιον της Επιτροπής Λίμπερ και να σα παρουσιάσω την πρόοδο του φορέα μα τον τελευταίο χρόνο. Πριν λάβω το λόγο, να πω κάτι για την εντολή μα, όπω είπε ο πρόεδρο μα, ο πρόεδρο σα. είμαστε αρμόδιοι για τη λειτουργή ε, διαχείριση του συστήματος για τις υποξενικές θεωρήσεις, το ΣΥΣ του Σέγγεν και του Eurodac και επίσης δίνουμε και εκπαίδευση για τους αρμόδιους από τα κάτι για τα συστήματα αυτά. Πέρσι ήταν ένα δύσκολο έτος για μας, είμαστε νέος φορέας και ο στόχος μας ήταν να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον οργανισμό αυτό και να αρχίσουμε τις λειτουργίες μας και συμφωνήσαμε φέτος με τους υπευθύνους των κρατών μελών στο Διοικητικό μας Συμβούλιο για τις προτεραιότητες που θα πρέπει να θεσπίσει ο φορέας μας. Η κεντρική στόχη λοιπόν του φορέα είναι η δημιουργία του οργανογράμματος μας, το να δημιουργήσουμε κέντρα αριστείας και επίσης το να κάνουμε εταιρικέ σχέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να αυξήσουμε την προσθέμενη αξία του φορέα μας προς τους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση λοιπόν με τα κύρια εγχειρήματά μας, θέλω να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής σας ότι υπάρχουμε με στόχο να μπορέσουμε μέσα, δημιουργήθεια για να πάρει μέσα σε 9 μήνες όλα τα εγχειρήματα που ε, πρέπει να διαχειρίζεται. Τώρα υπάρχουν οι κανονισμοί για τη διαχείριση των ασφαλών πληροφορικών δικτύων και όλα τα συμβούλια τα οποία είχαν προηγουμένως ε, συναυθεί σε σχέση με τη διαχείριση των συστημάτων αυτών έχουν μεταφερθεί στον φορέα μας και εμείς είμαστε αρμόδιοι για τη διαχείριση αυτών των ε, συμβάσεων. Ε, και για να καταλάβετε πώς λειτουργεί ο φορέας μας, εμείς αναλάβαμε και περαιτέρω καθήκοντα τα οποία δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα εργασίας μας πέρσι. Σε σχέση με τη δημιουργία <clears throat> μιας ε, δομής των φορέα μας υπάρχει το οργανόγραμμα το οποίο διαμορφώθηκε το 2013 επί τη βάση της αρχικής σχεδίασης, δηλαδή στο τέλος του 2013 είχαμε 120 υπαλλήλους στον φορέα μας, μεταξύ των οποίων και υπεύθυνη ασφαλείας, αρμόδιος ε, προστασίας δεδομένων και εσωτερικός ελεκτής. Επίσης πετύχαμε την δημοσιονομική αυτονομία στις 22 Μαΐου του 2013 εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου για να εξασφαλίσουμε την καλή διακυβέρνηση και τη σωστή οικονομική διαχείριση και τέλος, κάτι που είναι επίσης σημαντικό, υπήρξε συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο για τους στρατηγικούς μας στόχους και τις προτεραιότητες για το χρονικό διάστημα 2014-2020. Ο τρίτος τομέας προτεραιότητας να δημιουργήσουμε τα θεμέλια για κέντρα αριστείας, ετοιμάσαμε ένα πλαίσιο εσωτερικής διακυβέρνησης που ξεκίνησε η λειτουργία το 2013 και είναι εν εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία εσωτερικών υπηρεσιών όπως είναι η Επιτροπή για τον Προϋπολογισμό και τα Χρηματοοικονομικά, την ε, Επιτροπή Στατηγικού Σχεδιασμού που θα επιτρέψει μια σωστή λειτουργία του οργανισμού και την εκπλήρωση των προσδοκιών των εμπλεκομένων. Επίσης θα αναπτύξουμε και το εσωτερικό μοντέλο του φορέα ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματική λειτουργία, ακολουθώντας τα πρότυπα του κλάδου για τις, πληροφορίες τις τεχνολογίες πληροφορίας. και μετά από τα πρώτα αυτά βήματα έχουμε και ένα εταιρικό μητρό κινδύνου, το οποίο ενημερώνεται τακτικά ώστε να ξέρουμε ότι όλοι οι κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον ρόλο του φορέα μας βρίσκονται υπό διαχείριση. Έχει ξεκινήσει διαδικασία σχεδιασμού για το 2015 και έχει σχεδόν περατωθεί <clears throat> και επίσης υπάρχει ένας αναθεωρημένος ε, ένας ε, αναθεωρημένους κανονισμό λογαριασμών για την καλύτερη διαχείριση των λογαριασμών μας. Σε ό,τι αφορά τις εταιρικέ σχέσει, το 2013 ο φορέα μας ε, έχει συνάψει συμφωνίε βάσει μνημονίων ε, με την ε, ΣΥΠΟΛ και με την EU Home και έχουμε ήδη κοινέ ε, ενέργειες εκπαίδευση στα κράτη-μέλη. Έχουμε μνημόνιο κατανόηση με την Frontex και σχεδιάζουμε να κάνουμε από κοινού συγκεκριμένε δράσει που βρίσκονται στην αρμοδιότητα και των δύο αυτών φορέων. Έχουμε ένα κοινό μνημόνιο επίσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναμένουμε ότι θα υπογραφεί στους επόμενους μήνες και το οποίο βάσει του κανονισμού που θεσπίζει το φορέα μας προβλέπεται επίσης άρθρο 7 παράγωγος 2 και βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στις συμβουλευτικές μας ομάδες για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενώπιών μας. Εν κατακλείδη, το 2013 ήταν πολύ επιτυχές για το φορέα μας. Έχουμε ε, καλύψει τις προσδοκίες των εμπλεκομένων, έχουμε εκτελέσει πλήρως το πρόγραμμά μας και έχουμε δημιουργήσει στερεά ε, θεμέλια για την μελλοντική μας εργασία. Για τις προτεραιότητες του 2014. Το πρόγραμμα εργασίας και τα καθήκοντα του φορέα μας για το 2014 είναι εξελικτικού χαρακτήρα. Θα βασιστούν σε αυτά που έχουν επιτευχθεί ήδη το 2013 και οι τομείς προτεραιότητες που είχαν συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των κρατών μελών στο διοικητικό μας συμβούλιο δεν ποικίλουν από τις προτεραιότητες του 2013. Αλλά και πάλι ο φορέας μας θα συνεχίσει μια εξελικτική πορεία για την επέκταση των ενεργειών του, θα αναπτύξει και θα βελτιώσει την εσωτερική του διαχείριση και την δημοσιονομική διαχείριση και ιδίως την επίτευξη των προτεραιοτήτων. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει εξέλιξη των πληροφορικών συστημάτων για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι, ώστε να εξασφαλίσουμε και επίσης θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανονισμοί της Eurodax στο σύστημα το πληροφορικό και η συμβολή μας στην πρωτοβουλία για τα ΕΦΗ e, σύνορα είναι να δώσουμε ένα πιλωτικό σχέδιο για τα ευφυή σύνορα, ένα από τα κύρια λοιπόν στοιχεία της δραστηριότητά μας. Από την πλευρά της διακυβέρνησης έχουμε εγκρίνει μια μακροχρόνια στρατηγική, είναι η έγκριση του 2000, στρατηγικής 2014-2020 και τέλος μας ενδιαφέρει να υπάρξει μαζί με την ΣΥΠΟΛ της ικανότητάς μας να έχουμε καλύτερη τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και μας ενδιαφέρει να εκπαιδεύσουμε και να διατηρήσουμε το προσωπικό αυτό. Καταλήγοντας, πρέπει να πω ότι αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις εφέτος. Θα αντιμετωπίσουμε αυξανόμενες προσδοκίες και αιτήσει από τα κράτη-μέλη και τους άλλους εμπλεκόμενους αλλά είμαι σίγουρος ότι λόγω των σε θεμελίων που έχουμε δημιουργήσει το 2013, ο φορέας μας θα είναι πολύ επιτυχής για να μπορέσει και πάλι να ανταποκριθεί σε όλες τις προσδοκίες. Θα ήθελα να κλείσω λοιπόν και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την πρόοδο του φορέα μας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω οτιδήποτε ερωτήματα. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε και να ξεκινήσει η συζήτηση. Τώρα θέλει κανεί από τους συναδέλφου. Πολύ ωραία, ας ξεκινήσουμε. Όσοι θέλουν να κάνουν παρατήρηση. Και τον κύριο Κοέλιο. Τον ακόμα πρώτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μόλις έφτασα. Και ω εκ τούτου δεν έχω ακούσει την ομιλία του κύριου Καρκόφ. Αλλά ξέρω πολύ καλά την ε, δουλειά που κάνει. Στη Λίζα. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντική και καλή είναι η δουλειά που κάνει ο κύριος Γκαρκόφ με την ομάδα του. Ιδιαίτερα κάνουν καταπληκτική δουλειά, είτε πρόκειται για την Εστονία, είτε πρόκειται για το Στρασβούργο, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε κράτος μέλος ζητήσει την υποστήριξή τους. Και θέλω να πω ότι βλέπω όποτε ακούω τον κύριο Γκαρκόφ ότι είναι πολύ αισιόδοξο. Με όλες τις ε, περικοπές, τις δημοσιονομικές που προτείνει το Συμβούλιο, είναι αξιο, άξιο θαυμασμού το πόσο καλά δουλεύει η Λίζα, αλλά επίσης και πάνω απ' όλα πόσο αισιόδοξο είναι για το μέλλον ο κύριος Γκάρκοφ. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε μελλοντικέ δημοσιονομικές περιόδους, ώστε να μην περικόπτουν τα κονδύλια τόσο, ώστε να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ευχαριστώ κύριε Κοέλιο. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Θέλει κανείς άλλος μια παρατήρηση, άλλος βουλευτής. Well, Yeah. Απάντηση κύριε Γκαρκόφ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κύριε Κοέλιο. Ναι, είπα ότι θα έχει προκλήσει μεγάλες μπροστά τα επόμενα χρόνια η υπηρεσία μας αλλά ένα από τα ιδιαίτερα βήματα, ειδικά όταν μιλάμε για διακυβέρνηση, όταν μιλάμε για οικονομική διαχείριση, από τα βήματα και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε θα έχουν να κάνουν με την παραγωγή έργου με δεδομένες τις δημοσιονομικές ε, περικοπές, με τους περιορισμούς αυτούς. Προσπαθούμε λοιπόν να συνδυάσουμε τους βέλτιστους δυνατούς σπόρους, ανθρώπινους και οικονομικούς, ώστε να εξυπηρετήσουμε σωστά τις προτεραιότητες μας όταν έρχεται η ώρα. Είμαι, αν όχι αισιόδοξο πάντως αισθάνομαι ε, ότι μπορώ να διαβεβαιώσω με ασφάλεια πώς θα επιτελέσουμε το έργο μας σωστά και στα επόμενα χρόνια παρά τις περικοπές. Κύριε Γκάρκοφ, θέλετε να κάνετε ένα πρόσθετο σχόλιο στα όσα είπατε. ότι θα αρχίσετε να ασχολείστε με FEE σύνορα, με το σύστημα εφιών e σύνορων και ότι χρειάζονται οργανωτικοί πόροι για την ε, αποτελεσματική λειτουργία τέτοιου είδους συστήματος πληροφοριών και το σχετικό ε, μηχανισμό και βέβαια το νομικό πλαίσιο, την ένταξη στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απάντηση. Ναι, να κάνω πρώτα μία διευκρίνηση μια μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παραχθεί. Εμείς θα συμβάλλουμε ενεργά στην μελέτη αυτή ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες για το, σύστημα, για το σχεδιασμό του συστήματος. Το πρόγραμμα εργασίας ορίζει για φέτος την φάση προγραμματισμού των απαιτούμενων για την υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος των ευφυών συνόρων πόρων. Αυτό έχει προβλεφθεί εφόσον βέβαια προχωρήσει το νομικό πλαίσιο και εγκαθιδρυθεί το νομικό πλαίσιο. Εάν γίνει αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε το 2016. Αλλά δεν, προφανώς δεν μπορούμε όπως, όπως φαντάζεστε να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η νομική διαδικασία για να αρχίσουμε τη δουλειά εμείς από το 2016 και μετά. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει παράλληλα να ετοιμάσουμε τη νομική πρόταση και τη μελέτη, να συμβάλλουμε σε αυτά και βέβαια και στο πλαίσιο της Frontex εργαζόμαστε προκειμένου να προετοιμάσουμε και να ε, εξασφαλίσουμε τους πόρους που απαιτούνται, που επί τη ευκαιρία θα ήθελα να αναφέρω ότι καταγράφονται και στην ε, στον πολιετή σχεδιασμό για το προσωπικό της υπηρεσίας 2015-2017, ώστε να έχουμε την ορατότητα εκείνη των αναγκών που θα μας επιτρέψουν να συζητήσουμε την κατάλληλη ισορροπία με δεδομένη τη γενικότερη κατάσταση στον προϋπολογισμό και βέβαια τις ανάγκες σχέση με τις υπηρεσίες. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο, Λοιπόν, όσον αφορά την ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση που ακούσαμε, εκ μέρους του κ. Γκάρκοφ, θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Συμφωνείτε? Έτσι φαίνεται. Το επόμενο σημείο έχει προγραμματιστεί για τις 9.45. Ο κ. Προτεσίεβιτς είναι ο εισηγητής. Δεν είναι εδώ για την ώρα. Προτείνω λοιπόν διακοπή ενός τετάρτου. Εντάξει. Σε 15 λεπτά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. <laughs> shall λοιπόν, Να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε όπως προβλέπετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ενημερώθηκα ότι ο κύριος Προτασίεβιτς, ο εισηγητής μας για το προσεχές θέμα, δεν θα μπορέσει να έρθει. Ο ίδιος θα τον αντικαταστήσει όμως η κυρία Χιμένες Σερίλ, συνάδελφος. Θα συζητήσουμε πολύ μάτι τις τροπολογίες που έχουν τεθεί στο σχέδιο εκθέσεως και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την συζήτηση των τροπολογιών και την υποβολή της ε, γνωμοδότης νομικής επιτροπής για την έκθεση του κυρίου Πρωτασίβιτς για τις νέες ψυχότροπες ουσίες. Και βέβαια το θέμα των ελέγχων των τάξεω σε σχέση με τα στοιχεία τη αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων και τι ποινέ που ισχύουν στον τομέα τη παράνομη διακίνηση ε, ναρκωτικών κτλ. Έχουμε 127 και τροπολογίε για, για την έκθεση και 28 για την οδηγία. Θα ακούσουμε την κυρία Ισερή και μετά τους κοιόδες εφόσον το επιθυμούν. Νομίζω πρώτα απ' όλα κυρία Σερίλ πρέπει να ακούσουμε ποια είναι η γνωμοδότηση της νομικής, επιτρο... της νομικής υπηρεσίας, την οποία εδώ εκπροσωπεί ο κύριος Βισάτζο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, well, I think I... Νομίζω ότι μπορώ να είμαι σχετικά σύντομος. διότι διαπιστώνω ότι η ουσία τη γνωμοδότησή μα έχει ληφθεί υπόψη σε αρκετέ τροπολογίε, αλλά πρώτα απ' όλα ας μιλήσω για το γενικό πλαίσιο. Έχετε δύο προτάσει: Μία αφορά κανονισμό εσωτερική αγορά, που αφορά περιορισμούς ως προς την διάθεση στην αγορά ορισμένων ουσιών που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβείς και οι άλλοι οδηγία δυνάμει του άρθρου 23.1 της συνθήκης δηλαδή ε, νομοθέτημα του ποινικού δικαίου και που έχει να κάνει με την υλοποίηση επάφαση του 2004 και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιβάλλει ποινικές κυρώσεις σε ιανδήποτε εσκεμμένη παραβίαση των περιορισμών που ισχύουν σε σχέση με την εσωτερική αγορά, δυνάμει του κανονισμού εσωτερικής αγοράς. Και καλούμαστε λοιπόν να επαληθεύσουμε εάν υπάρχουν ζητήματα νομικού τύπου από το γεγονός ότι ο κανονισμός προβλέπει για τις προβλέπει για τις εξουσιοδότηση πράξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα λαμβάνονται εφόσον ε, ζητείται ζήτημα κυκλοφορίας επιβλαβών ουσιών και την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων δυνάμει της οδηγίας εφόσον παραβιαστούν αυτές οι απαγορεύσεις για τις απαγορευμένες ουσίες. Εμείς διαπιστώνουμε ότι το άρθρο 13 του Κανονισμού Εσωτερικής Αγοράς παρουσιάζει ζητήματα διότι ο κατάλογος των κριτηρίων με τα οποία ε, εντοπίζονται, καταγράφονται οι επικίνδυνες ουσίες ε, στην απόφαση επιτροπής δεν είναι εξαντλητικός. Πράγμα το οποίο δείχνει ιδιαίτερα ο όρος ιδίω in particular στον τίτλο του 13.1 στο κείμενο του 13.1 στο άρθρο 21 της συνθήκης μπορεί να εφαρμόζεται μόνο κάτι το οποίο, να, με εκτελεστική πράξη, μόνο κάτι το οποίο ήδη προβλέπεται στον κανονισμό ή την οδηγία. Εφόσον δεν είναι εξαντλητικός λοιπόν ο κατάλογος των κριτηρίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κάποιον τρόπο όταν ε, χαρακτηρίζει, εισάγει νέες ουσίες, εντοπίζει νέες ουσίες, κατά κάποιον τρόπο τροποποιεί το αρχικό νομοθέτημα. Βρίσκουμε λοιπόν διάφορες λύσεις να προτείνουμε για το ζήτημα αυτό, να προβλέπονται κάτι εξουσιοδότης συμπράξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορούν να υποκαταστήσουν τα κριτήρια αυτά, εφόσον θεωρηθεί σκόπιμο, ή να θεσπιστεί εξαντλητικός κλειστός κατάλογος του, κριτηρίου στο, του, των ε, κριτηρίων στο ίδιο το κείμενο, το νομοθετικό. Και επίσης η προτάσεις της Επιτροπής προβλέπουν, προβλέπεται ότι θα έχουν μια αυτόματη, διασύνδεση αναφορά στις ε, ουσίες που καταγράφονται δυνάμει του, της νομοθεσίας για την ιστορική αγορά, του ποινικού δικαίου για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή θα πρέπει τα κράτη-μέλη αυτομάτως να θεωρούν ποινικό αδίκημα ή αδίποτε διακίνηση ουσίας περιγράφεται σε αυτές τις αποφάσεις. Αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονό ότι θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει, να αναθεωρήσει το επίπεδο του κινδύνου του σχετικού με τι ελεγχόμενε ουσίε και ω εκ τούτου να τροποποιήσει τον, ε, την απόφαση. Και βλέπουμε ότι δεν είναι σαφέ από το κείμενο που καταθέτει η Επιτροπή το ότι και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υποχρεωθούν να βγάλουν την ουσία αυτή από το ποινικό τους ε, νομικό πλαίσιο την πονική του νομοθεσία και να σταματήσουν να επιβάλλουν κυρώσει σε περίπτωση διακίνηση τέτοιων ουσιών. Αυτά είναι τα δύο σημεία λοιπόν που εντοπίζουμε εμεί ως προβληματικά, νομοτεχνικά. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις μας και νομίζω ότι αυτά που είπα αρκούν. Πολύ ευχαριστώ να ακούσω ερωτήσει εφόσον χρειάζεται. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Βυζάντζο. Ακούσαμε την νομική τοποθέτηση. Ας παρουσιάσει η κυρία Χιμένα Φιχαρίλ τους τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, ελέγχθη, θα ασχοληθώ με τα θέματα των τροπολογιών, αυτά που μου ανέφερε ο κ. Ποστάσιεβιτς, ο οποίος βέβαια δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι επειδή μετά θα λάβω το λόγο για την αρμόδια οδηγία, εδώ είναι πολύ σαφής η απόψη του κυρίου Προτάσχευης για τις ε, τροπολογίες, αλλά αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις για τον κανονισμό, ε, απευθυνθείτε στον ίδιο ή στείλτε του email ή οτιδήποτε. Εγώ δεν είμαι αρμόδια για να αναφερθώ στα θέματα αυτά, μόνο για την οδηγία και τις τροπολογίες μπορώ εγώ να αναφερθώ. Έρχομαι λοιπόν σε αυτά που λέει ο κύριος Πορτάσιβιτς. Ε, υπάρχουν 104 τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί για τις νέες ψυχοτρόπες ε, ουσίες. Ο εισηγητής θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη της Επιτροπής για την εξισορροπημένη και πλήρη προσέγγιση τους και θέλει να υποστηρίξει το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων. Χαιρετίζει την τροπολογία που έχει τις τροπολογίες που διευκρινίσουν και αυξάνουν την νομική ασφάλεια αυτού του κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό επίσης θέλει να υποστηρίξει τις τροπολογίες του κύριου Χέντ στο, στα άρθρα 11, 12 αλλά και 13. Αυτό ισχύει και στις τροπολογίες που έχουν από τον κύριο Φιλίδη για τις αιτιολογικές σκέψεις. Σε ορισμένε από αυτές όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η διατύπωση συνάδει με την ε, επιχειρηματολογία για την εσωτερική αγορά. Ο κύριος Πορτασίβιτς επίσης δέχεται όλες τις τροπολογίες που τονίζουν το συμπληρωματικό χαρακτήρα του κανονισμού που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο λόγω των ιδιαίτερων συνδικών που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή πιο αυστηρών κανόνων από αυτούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζει επίσης την τροπολογία που ζητά τα προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευση κατά της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και επίσης τη στόχευση των ομάδων που βάσει των στοιχείων είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Όπως λένε τροπολογίες της κυρίας Ματιό και του κυρίου Πέρκελ, όπως και αυτές της, επιτροπή της Υποστήριζε και τι τροπολογίε που ζητούν μια πιο δυναμική και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών για τι ψυχοτρόπε ε, ουσίε για τι οποίε ο αρμόδιος φορέας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει καλύτερη πρόσβαση και να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως λέει η τροπολογία του κυρίου Σκούρια, του κυρίου Βέμπερ και του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Τούτο λεχθέντον όμως θα ήθελε να υπογραμμίσει και ορισμένε τροπολογίε που είναι για αυτόν προβληματικές. Δεν μπορεί να δεχτεί την τροπολογία του κυρίου Τριανταφυλλίδη για το άρθρο 6 σε σχέση με την κοινή έκθεση η οποία θα αποδυναμώσει το ρόλο της Ευρωπόλ στο προκατακτικό στάδιο της εκτίμησης του κινδύνου αυτών των ψυχοτροπικών ουσιών θεωρεί ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις ε, διαδικασίες που υπάρχουν και όχι να αλλάξουμε ένα εργαλείο το οποίο έχει λειτουργήσει σωστά. Και εξάλλου και οι δύο φορείς αντιμετωπίζουν διαφορετικές πηγές του κινδύνου που μπορεί να προκύψει από ψυχοτροπικές ουσίες, επομένως η συνεργασία τους θα πρέπει να είναι μια σωστή και αποτελεσματική βάση για την εκτίμηση κινδύνου που θα γίνεται από τις επιστημονικές επιτροπές μαζί με το φορέα για την παρακολούθηση των ναρκωτικών. Υπάρχει η τροπολογία του κυρίου Σκούρια στο άρθρο 11 που αναφέρεται στις νέες ψυχοτρόπες ουσίες για τις οποίες ο κύριος Κοτασιέβιτς κατανοεί με την επιχειρηματολογία αλλά θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση και δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής καμία λύση. Τέλος, υπάρχει ε, μεγάλη αντίδραση από τους σκιώδεις εισηγητές σε σχέση με τη χρήση κατεξουσιοδότηση πράξεων, κάτι το οποίο συμφωνεί και με τη θέση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για τα θέματα αυτά. Καταρχήν ο εισηγητής υποστηρίζει αντί για εφαρμοστικές πράξεις να είναι πράξεις κατεξουσιοδότηση, αλλά για τη σωστή λειτουργία αυτού του κανονισμού θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το να υπάρξει ένα ταχύς, μηχανισμός ταχείας αντίδρασης και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συστηθούν περισσότερο για να αποφύγουμε μια έγκριση αντιπαραγωγικών πρόνοιων. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με το άρθρο 9 για τις προσωρινούς περιορισμούς στην αγορά καταναλωτών όταν χρειάζεται μια ταχεία δράση της Κομισιόν λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρξουν σε αυτή σαφή κριτήρια, παραγωγικά θάνατοι και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή των, κατα... των εφαρμοστικών πράξεων <clears throat> είναι πιο αποτελεσματική κατά τον κύριο Προστάσεβιτς, αλλά είναι ανοιχτό σε περαιτέρω συζήτηση. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτό το τελευταίο σχόλιο και τώρα θα έρθω στο θέμα της δικής μου τροπολογίας. Και θα μιλήσω τώρα ισπανικά. Χωρίς μικρόφωνο, πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές οι οποίοι παρουσίασαν τροπολογίες για την οδηγία. Και αναφέρομαι τώρα στην οδηγία ως τον κανονισμό το μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών που έχουν παρουσιαστεί θεωρώ ότι εμπλουτίζει αυτή την έκθεση. Παρ' όλα αυτά έχω ορισμένα σημεία όπου θέλω να σταθώ. Η τροπολογία σε 7, 21 και 22 της κυρίας Head ε, έχουν σαν στόχο να δώσουν εξουσιοδότηση στην Κομισιόν για να τροποποιήσει το παράδειγμα μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων και όχι εκτελεστικό πράξεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη στην έκθεση. Η μόνη μου ανησυχία σχετικά είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχανισμό κατεπήγοντος σε περίπτωση μεγάλων κινδύνων για την υγεία για τις κατεξουσιοδότηση πράξη. Αν υπάρχουν όμως ε, κατεξουσιοδότηση πράξη στην τρέχουσα οδηγία, υπάρχει πάντα εναλλακτική λύση να γίνει αυτό στο άρθρο 13 του κανονισμού που αναφέρεται στους ε, σοβαρούς κινδύνους και τις προσωρινές ε, μορφές περιορισμού της αγοράς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το επιβεβαιώσει και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου σε σχέση με την ιατρική επισκόπηση. Αυτά δεν είναι θέματα αυτής της τρέχουσας οδηγίας, αλλά έχουν να κάνουν με, τις, με την οδηγία σε σχέση με τα φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν σαν στόχο την ανθρώπινη χρήση. Η τροπολογία της κυρίας Βέλτ στην 17 αναφέρεται σε μη ε, κερδοφόρες ε, χρήσης ε, ναρκωτικών, ότι πολλές φορές προσφέρονται ναρκωτικά τζάμπα για να προωθήσουν την τοξικομανία. Δεν συμφωνώ με αυτή την τροπολογία. Επίσης θέλω να πω ότι αυτή η οδηγία δεν αναφέρεται στον καταναλωτή ναρκωτικών. Αυτό αναφέρεται στην τροπολογία 3 της, ε, του σχεδίου έκθεσή μου, Επομένω δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να επαναλάβω κάτι το οποίο έχει γίνει σαφέ στην τροπολογία μου Μόνο τρία άλλε τροπολογίε όπω η 11, η 12, η 13, η 14 και η 18 εκφεύγουν <clears throat> του πεδίου εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Η πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τύχει επαρκού εναρμόνιση. Γι' αυτό πιστεύω ότι η αποδυνάμωση οποιασδήποτε ρήτρα στα θέματα αυτά δεν θα είναι θετική, τουλάχιστον στην τρέχουσα οδηγία. Εγώ προσωπικά προτιμώ να προωθήσω την, ε, το συντονισμό και τη συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ε, ουσιών. Στην τροπολογία 20, κύριος Βάτιμο θέλει να εξασφαλίσει ότι θα έχουν γίνει τα απαραίτητα εφαρμοστικά μέτρα στα καθημέρι δύο χρόνια μετά από την έκδοση αυτή τη οδηγία. Αλλά αυτό δεν είναι επαρκή χρόνο για να έχουμε αρκετέ πληροφορίε για να εξετάσουμε τα στοιχεία αυτά. Αυτό δεν, έχει, δεν σημαίνει ότι τα κρατη δεν πρέπει να δράσουν με οκίτητα για να αντιμετωπίσουν το εμπόριο ναρκωτικών. Τέλο, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιβάλλοντο, τη οποία οι τροπολογίε προ την κατεύθυνσή μα ήταν πάρα πολύ χρήσιμε. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μπεσερίλ. Ε, θα θέλαν τώρα οι σκιώδες να λάβουν το λόγο. Κύριε Χέντ, θέλετε να πείτε κάτι ως σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ την κυρία Μπεσέρη για την ε, παρουσίαση αυτή. Τι κρίμα που ο κύριος Προστασίεβιτς δεν μπορούσε να είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, αλλά έχω πάρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα ήθελα απλώς να εξηγήσω το νόημα των τροπολογιών μου, στις οποίες αναφέρθηκε η εισηγήτρια ένας μεγάλος αριθμός των τροπολογιών, έχουν να κάνουν με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη χρήση κατεξουσιοδότηση πράξεων θέλω να εξηγήσω ποια είναι η λογική αυτών των τροπολογιών και ελπίζω ότι και οι άλλες πολιτικές ομάδες θα τις υποστηρίξουν. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να υπάρχουν <clears throat> τροπολογίες στον κανονισμό τε και στην οδηγία που να κάνουν σαφές ότι τα κριτήρια για την αξιολόγηση του κινδύνου αν είναι υψηλό ή χαμηλό ο κίνδυνο, θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων σαφή. Εάν η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξει αυτή η ταξινόμηση, αυτό πρέπει να γίνει με κατεξουσιοδότηση πράξης. Αυτό θα εξασφαλίσει την ε, ε, σαφήνεια δικαίου και την ασφάλεια δικαίου και το ρόλο του Κοινοβουλίου. Για την οδηγία έχω την τροπολογία 1 που αφορά τις αποφάσεις για ποινική δίωξη όπου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλέκεται ως νομοθέτης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου. Επίσης έχω εξετάσει την εισαγωγική παραδοσίαση της Κομισιόν. Δεν ε, ξέρω αν κατάλαβα λάθος, αλλά <clears throat> νομίζω ότι αναφερθήκατε στη δυνατότητα των κρατών μελών να προχωρήσουν σε πιο αυστηρές ρυθμίσεις σε σχέση με τη ρύθμιση των ε, ναρκωτικών ουσίων. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που θέλουν πράγματι να πράξουν τα κράτη-μέλη και αν δεν πρέπει να παραμείνει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κατάλαβα τι είπε η Κομισιόν. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το είχαμε συζητήσει ήδη. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Χέντ. Κάποιος άλλος. Ο κύριος Μπρόγκς. Κύριε Μπρόγκς έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σαν φάσμα είμαι, δεν είμαι σκία. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν για το πρόβλημα από αυτά που προτείνονται. Ο εντοπισμός του προβλήματος είναι ευκολότερος από τη λύση. Υπάρχουν ουσίες που δεν καλύπτονται από το ποινικό δίκαιο και που χρησιμοποιούν οι νέοι και υποφέρουν από αλλαγέ όσον αφορά τη συνείδηση, συμπεριφορά, αντίληψη, αλλάζει η συμπεριφορά του και ίσω να είναι μακροπρόθεσμε οι αρνητικέ συνέπειε. Ποια είναι η δυσκολία, ότι η ταυτότητα των ουσιών και η ονομασία των ουσιών, αν όχι όταν συστατικά, συνεχώ αλλάζουν. Οπότε προλαμβάνουν, προηγούνται τη νομοθεσία. Αποκρυφά εργαστήρια, σαν αδίουσες Οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία ε, παράγονται αυτές τις ουσίες που εκεί δεν υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον έλεγχο της παραγωγής. Έτσι λέει η έκθεση. Λίγο ηρωνικό το βλέπω στην περίπτωση της Κίνας. Δηλαδή μπορούν να καταστήλουν την αντιπολίτευση και τους αντιφρονούντες, αλλά δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις επιβλαβείς οικονομικές δραστηριότητες. Και κάτι άλλο ελληνικό. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με αυτές τις χώρες. Δεν ξέρω μέσω οποίων διάβλων συνάπτουν συμφωνίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει από την άλλη ότι πρόκειται περί διεθνού προβλήματο. Σωστό αυτό. Άρα χρειάζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω λύση. Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ένωση αυτέ οι λέξει δεν είναι κάτι συνώνυμο. Παγκόσμια προβλήματα απαιτούν παγκοσμίου επίπεδου λύσει. Αυτέ παράγονται μόνο μέσω διεθνών συνθήκων. Με το μέγιστο αριθμό υπογραφών. Όχι μόνο υπογραφέ 28 χωρών. Στην έκθεση εκφράζεται ανησυχία του Δηλαδή ότι οι δράσει των μεμονωμένων κατών μελών για την επίλυση του προβλήματο ίσω απειλήσουν την ενιαία αγορά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ανησυχητικό σχόλιο. Αυτό φαίνεται να μα ανησυχεί τελικά. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το άνοιγμα των συνόρων δημιούργησε ενιαία αγορά. Όχι μόνο στα νόμιμα αγαθά, αλλά και σε όλα τα παράνομα αγαθά υπηρεσίε και του καρπού παρανόμων δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Μπρόξ. Υπάρχει σχόλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Προεδρία, μήπω θέλει να μας πει κάτι όσον αφορά τις τροπολογίες. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σπινούντ, η κυρία Σπινούντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Χιμένες και τον κύριο Μπρόν για τις σκέψεις που εκφράσαν για το πακέτο για τις ψυχότροπες ουσίες. Καλωσορίζω τις δύο των εισηγητών. Είναι πολύ επικοδομητικές. Θα βοηθήσουν να παγιωθεί το προτινόμενο σύστημα για να αντιμετωπίσουμε τις ψυχότροπες ουσίες. Θεωρούμε επίσης τις υποβληθήσεις τροπολογίες των μελών άκρως επικοδομητικές Βρίθουν ιδεών για τη βελτίωση των προτινομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τροφή προσκέψη. Θα τις εξετάσουμε διεξοδικά. Μπορούμε να πούμε ήδη ότι πολλές από αυτές θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο, δηλαδή βελτίωση της ταχύτητας και την αποτελεσματικότητα του συστήματος για την καταπολέμηση των ψυχότροπων ουσιών και θα μας βοηθήσουν να διευκρινίσουμε τη διάδραση μεταξύ εθνικών προσπαθειών και δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνουμε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χρήση εφαρμοστικών πράξεων και καταξουσιοδότηση πράξεων. Επαναλαμβάνω, για ποιους λόγους πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμοστική πράξη συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι προτείνουμε σαφή κριτήρια βάσει των κριτηρίων θα πρέπει ε, να δράζονται υποφάσεις για τα περιοριστικά μέτρα. Θα το εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα. Θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να βρεθεί η σωστή λύση για όλα τα προβλήματα που ετέθησαν από τους συζητητές. Καθώς και αυτά τα προβλήματα που αναφέρονται στις τροπολογίες, ευχαριστούμε πολύ για την επικοδομητική συνεργασία όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα μας βοηθήσει η στάση αυτή να πετύχουμε γρήγορα συμφωνία τόσο ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπινόντ. Η ελληνική προεδρία, η κυρία Ραπτάρχη, έχετε το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, από την τελευταία ενημέρωση της Προεδρίας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, 23 ε, Ιανουαρίου, το Συμβούλιο, ε, σε πλαίσιο συνεδρίασης της Οριζόντιας Ομάδας Ναρκωτικών, εξέτασε, εξέτασε την πρόταση του κανονισμού κατά δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις του, 6 και 7 Φεβρουαρίου. Προεδρία κατά την πρώτη μέρα της συνεδρίασης, 6 Δευτέρου, παρουσίασε αναθεωρημένη έκδοση ανωτέρου κανονισμού για ε, τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες για τα κεφάλαια 1, 2 και 3 και τα άρθρα 1 έως 13 σε αναθεωρημένο κείμενο συμπεριλήφθησαν βάσει προτάσεων της προεδρίας σχόλια των κρατών μελών σχόλια της επιτροπής ΛΥΜΠΕ καθώς και προτάσεις της κομισιόν και της νομικής υπηρεσίας του συμβουλίου. η συζήτηση διαμορφώθηκε σε δύο μέρη. σε πρώτο μέρος συνεχίστηκε η πρώτη ανάγνωση του κειμένου για τα κεφάλαια 4, 5 και 6 με αναλυτική παρουσίαση σχετικών άρθρων και σχολιασμό κρατών μελών ενώ στο δεύτερο μέρος ξεκίνησε η εξέταση στη δεύτερη ανάγνωση του κεφαλαίου 1 και 2, τα άρθρα 1 και 2, σε αναθεωρημένο έγγραφο. Η Προεδρία κάλεσε τα κράτη-μέλη, όπως αποστείλουν γραπτός προτάσεις για επαναδιατύπωση συναφών σημείων, με προτινόμενες προσθήκες, έως 20 Φεβρουαρίου, προκειμένου αναθεωρημένη έκδοση σχετικού εγγράφου, κοινοποιηθεί σε κράτη-μέλη προ προσεχού συνεδρίασης ομάδας εργασίας. Συμπερασματικώς μπορούμε να πούμε ότι εργασίες εξέτασης πρότασης του κανονισμού προχωρούν ε, και η Προεδρία προτίθεται να συνεχίσει να ενημερώνει την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ επί της προόδου των εργασιών, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προσεχή συνάντηση αρμόδιας ομάδας εργασίας του Συμβουλίου προβλέπεται να συνεδριάσει 27 ε, Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Καλώς κύριε Ραφτάκη. Έχοντας ακούσει λοιπόν την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν δεν έχετε άλλα σχόλια, μπορούμε να δώσουμε ξανά το λόγο στους ε, εισηγητές. Η κυρία Χιμένας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους σκιώδες εισηγητές και όλους τους άλλους βουλευτές που κατέθεσαν τροπολογίες και με τον τρόπο αυτό έχουν ε, διευκρινίσει και βελτιώσει πολλά σημεία της οδηγίας και του κανονισμού και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν η οποία έλαβε υπόψη την τροπολογία της κυρίας Χερτ που και εγώ είχα υποστηρίξει σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και επίσης ευχαριστώ και την νομική υπηρεσία για την διαθεσιμότητα να σε αυτήν τη συμφωνία και όπως είπα και προηγουμένως τονίζουμε ότι θέλουμε να έχουμε κατεξουσιοδότηση πράξη και όχι κατεκτελεστικές ε, πράξεις και βασίζομαι και στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για το θέμα αυτό για την οδηγία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και το Συμβούλιο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις συνεδρίες 27 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ κύριε Χιμένες. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε κοινή συζήτηση. Το σημείο 9 και το σημείο 10 αφορούν Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ενώση Αζερμπαϊτζάν για την επανειστοχή προσώπων που διαμένουν χωρί άδεια και σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Μαρία Γκαμπριέλ. Ας ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση της όλης καταστάσεως όσον αφορά τις συμφωνίες. Ξέρουμε ότι πάνε χέρι με χέρι και το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει σύμφωνη γνώμη πριν τεθούν σε σχέση συμφωνίες. Ας ακούσουμε λοιπόν την κυρία Γκαμπριέλ και μετά κάποιους σκιώδεις συζητητές. Κυρία Γκαμπριέλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την απόφασή της τη σχετική με τις συμφωνίες επανειστοχής και απλούστευσης έκδοσης θεωρήσεων με την Δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν. Για να γίνει μια, ή πριν να γίνει μια ε, σωστή παρουσίαση των εκθέσεων. Πρέπει κανείς να γνωρίζει καλά την κατάσταση. 30 Ιανουαρίου λοιπόν του 2014 στην Επιτροπή Λίβη είχαμε την ευκαιρία για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία απεδείχθη επικοδομητική και μας επέτρεψε να προχωρήσουμε στη δουλειά μας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ελήφθη υπόψη όπως άλλωστε και η γνωμοδότηση που μας απέστειλε η Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων και που έχει επίσης εγκριθεί. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω σήμερα την διαδικαστική αλλά και την πολιτική σημασία αυτής της εκθέσεως. Έχουμε καταρχάς την διαδικαστική της σημασίας προς τις διατυπώσεις δηλαδή και είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να εγκριθούν δύο συστάσεις με τις νέες συμφωνίες εισάγονται νέοι κανόνες χάρη στους οποίους απλουστεύονται οι ε, διαδικασίες και κάθεται πιο ταχείες και για την πολιτική σημασία ξέρουμε ότι οι δύο αυτές εκθέσεις προκύπτουν ως ε, αποτέλεσμα, ως ε, προϊόν της ε, ηθελημένης προσέγγισης και αποφασιστικής προσέγγισης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερβαϊτζάν. Επομένως θέλουμε να υπάρξει αυτή η προόδος ώστε να επαληθεύεται η βούληση για πολιτική ε, υποστήριξη της ελευθερίας διακίνησης των προσώπων μεταξύ των δύο πλευρών. Πιστεύουμε λοιπόν πρέπει να εμβαθύνουμε τις ε, ε, σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερβαϊτζάν ώστε να ανοίξουν τα σύνορα του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας. Θα αποτελέσει αυτό μια αναμφισβήτητη πρόοδο στον χώρο της κινητικότητας για τις τεχνικές διατυπώσεις της συμφωνίας για τη διευκόλυνση Θεωρητή διαβατηρίων. Έχουμε καταρχάς κάποια σημεία ότι θα περιοριστεί στα 10, στις 10 ημέρες η διαδικασία για την χορήγηση, για την απάντηση στην αίτηση ή μάλιστα σε περίπτωση δύο ε, επιτυχημένων διαδικασιών θα περιοριστεί στις 2 ημέρες ή μπορεί σε περίπτωση άκρος εξαιρετική να φτάσει μέχρι τις 30 ημέρες. Θα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες ετούντων, οι έχοντες ε, οι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων δεν θα απαιτείται να ζητούν ε, βίζα για σύντομη διάρκεια παραμονής. 35 ευρώ θα είναι το τέλος για τη θεώρηση, ορισμένοι θα απαλλάσσονται πλήρως του τέλους αυτού και προβλέπονται επίσης για τη χορήγηση θεωρήσεως πολλαπλών εισόδων ειδικέ διατάξεις, παραδείγματι ομάδες αξιωματούχων και οικογένειες αυτών. Για τη δεύτερη περίπτωση, τη συμφωνία της επανεισδοχής, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση της επανεισδοχής έχουν προσδοριστεί κανόνες με τη βάση της απόλυτης αμοιβαιότητας, Επίσης ε, προτείνεται από την αρχή η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας να γίνεται κατά τρόπον ώστε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ορίζονται οι τεχνικές πτυχές της διαδικασίας ε, και ένας κατάλογος μέτρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της συμφωνίας επανεισδοχής, τεχνικές διατυπώσεις δηλαδή, επιταχυμένες διαδικασίες, ε, τμήμα που έχει να κάνει με την διέλευση, το transit, την εφαρμογή των κανόνων σε διάφορες κατηγορίες ατόμων, πρώην, ε, ε, πρώην ε, κατοίκων, υπηκών καλύτερα που δεν έχουν λάβει υπηκότητα κράτους μέλους, που έχουν χάσει την ηθαγένεια από το Αζερβαϊτζάν, ατόμα που έχουν ενταχθεί παράνομα στο κράτος αίτησης, ενώ έχουν διέλθει από το κράτος προέλευσης, προσώης η αίτηση καλύτερα και ούτω καθεξής. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι στις δύο αυτές συμφωνίες λαμβάνονται υπόψη και ιδιαίτερε καταστάσεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και το Βασίλειο της Δανίας. Ως εισηγήτρια επίσης, πολύ ευχαρίστω να ακούσω παρατηρήσεις, συστάσεις, υποδείξεις των συναδέλφων, του οποίους προκαταβολικά και ευχαριστώ. Επισημένω δε ότι και οι δύο συμφωνίες ε, προβλέπουν την σύσταση, την ίδρυση μεικτών επιτροπών διαχείρισης που θα παρακολουθούν την απρόσκοπτη λειτουργία των συμβάσεων με συμμετοχή εκπροσώπων της Δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εκπροσώπηση και στις δύο περιπτώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών. Στην εκθέση, εκθέσεις απευθύνω σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επανεξέταση της σύνθεσης των μεικτών επιτροπών διαχείριση για μελλοντικέ συμβάσει, ώστε να συμμετέχει ευρύτερα αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιλαμβανόμενοι όμω πάντω και τα όρια αυτή τη συστάσεω και πάντω και στι δύο ε, περιπτώσει καλό την Επιτροπή να ενημερώνει σε κάθε στάδιο της ε, θέση εφαρμογή των συμφωνιών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικαλούμενη την απλή αρχή της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους για το χρονοδιάγραμμα, για την κατάσταση τροπολογιών προβλέπεται προθεσμία έως 18 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, αλλά με, με τον προσδορισμό ότι μόνο διαδικαστικού χαρακτήρα τροπολογίες είναι παραδεκτές και 20 Φεβρουαρίου έχουμε την έγκριση στην Επιτροπή των πολιτικών ελευθεριών. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία, την καλή συνεργασία για την έκθεση αυτή, όπω έχουμε άλλωστε ξεκινήσει από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και περιμένω εδώ να ακούσω τι θέσει των συναδέλφων από τι διάφορε πολιτικέ ομάδε, ώστε η ε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου να διαμορφωθεί με τα λόγου γνώσεως και πάνω απ' όλα με ένα ισχυρό μήνυμα που και διαδικαστικά θα αποσταλεί ώστε να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το Αζερβαϊτζάν κατά τρόπο αποφασιστικό γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκαμπριέλ. Λοιπόν, ακούσουμε τι έχουν να πούνε σκιώδεις. Η κυρία Τανόκα. Θέλετε να μιλήσετε. Έχετε το λόγο, κύριε Τανόκα. Ευχαριστώ. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας, τη Μαρία Γκαμπριέλ, για την έκθεση. Η ομάδα των Πρασίνων είναι υπέρ της διευκολύνσεως του καθεστώτος θεωρήσεων είναι θέση μας επί της αρχής. Όσον αφορά το Τζερμπαϊτζάν, υπογραμμίσαμε την ανάγκη να διοργανωθεί διαδικασία συμφωνίας, σύναυση συμφωνίας για διευκόλυνση των θεωρήσεων. Με την ίδια ταχύτητα θέλουμε να γίνει αυτό και ταυτόχρονα με τις συμφωνίες με άλλους ανατολικούς εταίρους μας. Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, το ξέρετε. Όσον αφορά την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, διαφορετικά ήταν η εξέλιξη, διαφορετική εξέλιξη. Συμφωνήσαμε πιο νωρίς με την Αρμενία από ότι με το Αζερβαϊτζάν και η ομάδα μας πρότεινε να κινηθούμε ταυτόχρονα. Δεν έγινε αυτό. Τώρα όμως είμαστε ικανοποιημένοι που η συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν είναι πρώτων θυρών και καλωσορίζουμε, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες όλων εκείνων που συνέβαλαν στην σύναψη συμφωνίας. Το θέμα της συμφωνίας επανεισδοχής είναι ένα άλλο ζήτημα. Βασική μας αρχή είναι ότι είμαστε κατά ερεσιμότητας όσον αφορά τις δύο συμφωνίες κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν ε, επικρατεί σύγχυση αβεβαιότητες σε κάποιες περιοχές υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την ηθαγένεια ανθρώπων ε, σε αυτές τις περιοχές Υπάρχει κάποιος κίνδυνος λοιπόν όσον αφορά τις ατομικές ελευθερίες και την ασφάλεια των ανθρώπων που θα καλύπτονται από τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Η ομάδα μας λοιπόν δεν υποστηρίζει τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντάνοκα. Άλλος που θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Μπρόντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρθηκε η φράση άτομα χωρίς έγκριση διαμονής. Αυτό είναι ένας εφημισμός όπως και η μη σε κανονικό επίπεδο μετανάστες. Φαίνεται ισορροπημένη αυτή η συμφωνία αλλά είναι απόλυτα μονόπαντη. Εγώ δεν μπορώ να βρω λοιπόν πώς θα το ονόμαζα αυτό το, αυτή τη συμφωνία, αλλά τέτοιες συμφωνίες είναι ε, παραδείγματα αυτής τη λογικής. Καταρχήν για την επανειστοχή όταν τα άτομα τα οποία βρισκόνται παράνομα σε μια άλλη χώρα πρέπει να γίνουν δεκτοί στη χώρα από την οποία προήλθαν. Αυτή είναι μια αμφίδρομη συμφωνία που εφαρμόζεται και στις δύο χώρες και στους πολίτες τους ή αυτούς που δεν είναι πολίτες της με μία μονάχα έλλειψη ισορροπίας. Μπορεί να υπάρχουν πιο πολλοί πολίτες του Αζερβαϊτζάν που ζουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι Ευρωπαίοι που ζουν παράνομα στο Αζερβαϊτζάν. Ένα άλλο μικρό πρόβλημα είναι ότι είναι υποχρεωμένες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεχτούν και πάλι πίσω τους πολίτες τους και αυτούς οι οποίοι έχουν απεκτηθεί την ε, υπηκότητά τους και αυτό θα πρέπει να το κάνει το Αζερβαϊτσάν για να μπορούν και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρει πίσω τους πολίτες, τους, πολίτες που μπήκανε μέσα στο Αζερβαϊτζάν για να αγοράσουν, να αποκομίσουν ορισμένα μανάτ σε επιδόματα κοινωνικής ασφάλειας εκεί. Επίσης υπάρχει το θέμα της φιλελευθερωποίησης στις προξενικές θεωρίες που είναι και αυτό αμοιβαίο. Οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να πάνε στο Αζερμπαϊτζάν με απλοποιημένε διαδικασίε και θα έχουν τη διαδικασία να μείνουν εκεί πέρα πέρα από το όριο τη βίζα παράνομα. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κανένα λογικό άνθρωπο που να θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και οι πολίτε του Αζερμπαϊτζάν θα μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα με την ίδια ευκολία και να γυρίσουν όταν θέλουν ή όταν του καπνίσει. Όλα αυτά δεν μου φαίνονται ιδιαίτερα αμοιβαία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε η Κομισιόν, η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου, ο κ. Νίλς Κόλμα είναι εκπρόσωπος της Κομισιόν από ό,τι γνωρίζω. Θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για τα σχόλιά του. Η έκθεση αυτή είναι κατά την άποψη της Κομισιόν ιδιαίτερα θετική και καλόδεκτη. Έχουμε κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις και κάποιες ε, διορθώσεις σε θέματα ουσίας που θα δώσουμε χωριστά στην εισηγήτρια για να τις ε, λάβει υπόψη της. Η έκθεση σωστά υπογραμμίζει ότι βρισκόμαστε εδώ στο ευρύτερο πλαίσιο της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης και έχει δημιουργηθεί, έχει αποφασιστεί να δημιουργηθεί το πλαίσιο για διακίνηση χωρίς προξενικές θεωρήσεις για τα μέλη αυτής της εταιρικής σχέσης και γι' αυτό αυτή η συμφωνία είναι ένα πρώτο βήμα. Οι δύο αυτές συμφωνίες είναι συνδεδεμένες γιατί φυσικά είναι σημαντικό να διευκολύνουμε την κινητικότητα με έναν τρόπο που θα είναι ασφαλής και γι' αυτό υπάρχει και η Συμφωνία Πενισδοχής που αποκτά την πλήρη σημασία της. Με αυτά τα πρώτα βήματα λοιπόν έχουμε πετύχει κάτι που είναι σημαντικό για τους πολίτες του Αζερμπαϊτζάν και το Αζερμπαϊτζάν είναι να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία και να τεθούν σε εφαρμογή αυτές τις συνδίκες το ταχύτερο δυνατό από αυτή την άποψη. Οι συστάσεις της εισηγήτριας να εγκρίνουμε αυτές τις ε, πρόνοιες είναι απόλυτα καλόδεκτη. Για τη συμφωνία τώρα επανεισδοχής, η έκθεση έχει όλες τις λεπτομέρειες, αυτή είναι μια συμφωνία πλήρους εμβέλεια αναφέρει όλες τις υποχρεώσεις και όλες τις απαραίτητε διαδικασίε για να μπορεί να υπάρξει καθημερινή λειτουργία αυτής της συμφωνία για τα κάτι μέλη μα και για τις αρχέ του Αζερβαϊτζάν. και υπάρχουν όλες αυτές οι εγγύησεις που εξασφαλίζουν ότι δεν θα γυρίσει κανείς στο Αζερβαϊτζάν αν κινδυνεύει με οποιοδήποτε τρόπο για τη συγκεκριμένη τώρα σύσταση του να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κοινή Επιτροπή Επανεισδοχής. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, ένα θεσμικό θέμα όπου η νομική μας υπηρεσία θα πρέπει να δώσει μια πιο συγκεκριμένη γνωμοδότηση από πλευρά πολιτικής όμως είναι ένα τεχνικό σώμα το οποίο κάνει συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομεριακές συζητήσεις για την εφαρμογή των συμφωνιών και δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και γι' αυτό κατά τη δική μας άποψη θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην σωστή πληροφόρηση του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή όχι μόνο αυτής της συμφωνίας αλλά όλων των συμφωνιών επανεισδοχής που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ήδη στόχος μας να το κάνουμε και προσβλέπουμε σε περαιτέρω βελτίωση αυτής της συνεργασίας. Σας ευχαριστώ και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία διευκόλυνσης προξενικών θεωρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο έτερος εκπρόσωπος της Επιτροπής, κύριος Πάλμαν, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για τη θετική έκθεση. Όπως είπε και ο συνάδελφος, είναι σημαντικές αυτές οι συμφωνίες για τις σχέσεις μας με το Αζερβαϊτζάν και γενικότερα το πλαίσιο της Ανατολικής Γειτονίας. Επομένως, καλωσορίζουμε αυτή τη θετική έκθεση. Δύο θέματα προέκυψαν, τα οποία, στα οποία θα απαντήσω πολύ στοματά. Αρχάς, δυνατότητα για συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μεκτή Επιτροπή εγώ προσυπογράφω πλήρως τις ε, θέσεις που εξέφρασε για το θέμα αυτό ο συνάδελφος από την ε, θέση της επανεισδοχής. Την πλευρά της επανεισδοχής είναι θεσμικά ζητήματα, είναι τεχνικές επιτροπές και στο άρθρο αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το Κοινοβούλιο, την ε, Ένωση, την εκπροσωπεί Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν βλέπω λοιπόν χώρο και περιθώριο για συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τέτοιου επιτροπές. Ασφαλώς όμως, όπως είπε και ο συνάδελφος, ενημέρωση για τα όσα θα ε, διαμείβονται σε αυτές τις επιτροπές που θα είναι πολυτεχνικού χαρακτήρα θα ε, απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για το έτερο ζήτημα και την παρατήρηση του κυρίου Βουλευτού για την ε, παραμονή ή μάλλον για την παρουσία υπηκόν του Αζερβαϊτζάν σε κράτη του χώρου Σέγγεν. δεν θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για διαδικασία απα, από την υποχρέωση θεώρηση, αλλά διευκόλυνσης. Και άρα θα έχουμε βραχυπρόθεσμες, βραχυχρόνιες θεωρίες διαβατηρίων, με περιορισμένη δηλαδή διάρκεια παραμονής. Εάν κανείς παραμείνει περισσότερο από ό,τι προβλέπεται στη θεώρησή του, τότε τίθεται σε λειτουργία η συμφωνία περί επανεισδοχής και ε, θα πρέπει να αποχωρήσει εφόσον έχει ενταχθεί παράνομα στο χώρο του, έχει σαχθεί παράνομα στο χώρο του Σέγγεν ή έχει ε, παραμείνει για διάστημα μεγαλύτερο από όσο το επιτρέπει η θεώρηση διαβατήριων. Ευχαριστώ πολύ για τις ετικέ εκθέσεις και με στη θέση σας έτερος για την ε, για τις συμφωνίες αυτές, κυρία Τομάνσκα, όχι. Η ελληνική προεδρία τότε παρακαλώ, αν θέλει να κάνει μια παρατήρηση, δήλωση, να συμβάλλει στη συζήτηση, όχι. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Ευχαριστώ και ξαναρωτώ την ε, κυρία Μαρία Γκαμπριέλη αν θέλει να κάνει κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τις παρεμβάσεις τους. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την θετική αντιμετώπιση εκθέσεως και ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις που δόθηκαν όσον αφορά τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, όσον αφορά τις εργασίες της Μικτής Επιτροπής. Καταλαβαίνω απόλυτα τα όρια της προτάσεως, καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι θεσμικό ζήτημα, αλλά επαναλαμβάνω την ιδέα που αναφέρθηκε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται περαιτέρω προβληματισμό όσον αφορά τη δυνατότητα πληροφοριών, όσον αφορά αυτά που συμβαίνουν στι τεχνικέ επιτροπέ και να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για την καλή συνεργασία, το διάλογο και ενθαρρύνω τους συναδέλφους ε, να κινηθούμε για να προχωρήσουμε γρήγορα στο θέμα αυτό, διότι είδαμε ότι είναι σημαντικό θέμα για την ευάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκαμπριέλ για την παρουσίαση των εκθέσεων. Αυτά για την ώρα. Πάμε στο επόμενο σημείο και πάλι κοινή συζήτηση που διεξάγεται έχουμε σημεία σχετικά το 11, το 12 και το 13, το 14 με τον ίδιο στόχο Αποφορά το σχέδιο εκθέσεως για ρύθμιση με την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά στο τομέα συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο, ίδιες ρυθμίσεις με τη Δημοκρατία τη Ισλανδία ρύθμιση με το βασίλειο της Νορβηγίας, παρομοίως με το πριγκιπάτο του Λίχτενστάιν. Ας ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση του σχεδίων εκθέσεως, λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις ρυθμίσεις εντάσσονται στη διαδικασία συμφώνου γνώμης. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του πριν τεθούσε ισχύ. Το λόγο έχει ο λόγο η κυρία Μετσόλα για να παρουσιάσει το σχέδιο συστάσεως, το σχέδιο εκθέσεως και μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Προεδρία. Κύριε Μετσόλα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, μπορεί να παίξουμε... Ε, λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, για να βοηθήσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη το άσυλο. Λοιπόν, το άρθρο 49 του κανονισμού της Υπηρεσίας διαθετεί, αναφέρεται ότι θα γίνουν ρυθμίσεις που θα καθορίζουν συγκεκριμένα τη φύση, το βαθμό, το πεδίο εφαρμογή και τον τρόπο με τον οποίο η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λίχτενστάιν θα συμμετάσχουν στι εργασίε ε, του Γραφείου Υποστήριξη. Η συμμετοχή των εν λόγω συνδεδεμένων χωρών στην υποστήριξη ε, θα είναι μια σημαντική διάσταση στο ρόλο της ΕΑΣΑ σύμφωνα με τον κανονισμό που δημιουργεί την υπηρεσία θα γίνεται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών και της ΕΑΖΟ που πιστεύω ότι θα ωφελήσει όλους μας. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, αυτά τα θέματα αποφασίζονται στα πλαίσια της Συμφώνου Γνώμης σχετικής διαδικασίας και έχω την πεποίθηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να δώσει σύμφωνη γνώμη του όσον αφορά τη διεκπαιρέωση των υποθέσεων αυτών, όσον αφορά τη συμμετοχή των χωρών στην Ευρωπαϊκή ε, υπηρεσία υποστήριξη για το άσυλο. Ταχύτερο δυνατόν προσβλέπω και σε συνεργασία με του σκιώδει όσον αφορά τα συγκεκριμένα αυτά θέματα. Όμω, και εδώ θέλω να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά την Ελβετία. Θα ήταν χρησιμότατο να έχουμε κάποιε διευκρινήσει όσον αφορά το πρόσφατο δημοψήφισμα και τα αποτελέσματα αυτού και να καταλάβουμε οι εσδήποτε ε, συνέπειε που θα έχει το αποτέλεσμα δημοψηφίσματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Ελβετία και προσβλέπω σε απόψεις για τη συγκεκριμένη έκθεση των συναδέλφων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ματσόλα. Λοιπόν, να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Μωράης, τον σκιώδη μας. Θα τα πάτε πρώτος, να πάρετε το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η Σκιώδης από τη δική μου πολιτική ομάδα δυστυχώ δεν μπορεί να είναι παρούσα, γι' αυτό θα πω ορισμένα λόγια εξ ονόματό τη, εάν δεν έχετε αντίληση. Η συμμετοχή των χωρών αυτών στο έργο της ΙΙΑΣ είναι προφανώς ένα λογικό βήμα διότι συμμετέχουν και στο σύστημα του Δουβλίνου και ευνοούν και την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης ε, και εξασφαλίζουν την καλύτερη ανάλυση και την πρώιμη προειδοποίηση για το Γραφείο Υποστήριξης του Συστήματος Ασύλου. Έχουμε ήδη λοιπόν πολύ χρήσιμε πληροφορίε που έχουν προέλθει από αυτή τη διαδικασία. Ο στόχο μα είναι να υποστηρίξουμε πλήρω το ρόλο αυτού του φορέα. Οι επιλογέ που ακούσαμε βέβαια ότι έγιναν από τους Ελβετούς θα έχουν χωρίς αμφιβολία κάποιες επιπτώσεις στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας. Και ίσως και η νομική υπηρεσία θα μπορέσει να μας δώσει και κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τον αντίκτυπο αυτής της πρόσφατης απόφασης που ελήφθη στο δημοψήφισμα της Ελβετίας σε σχέση με, την, με τον τρόπο που θα πρέπει να γίνει η συμμετοχή της Ελβετίας στο γραφείο αυτό υποστήριξης του συστήματος ασύλου. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή προσοχή για τη δυνατότητα αναστολής των διαπραγματεύσεων, αλλά προηγουμένως φυσικά θα πρέπει να ακούσουμε τα επιχειρήματα και της άλλης πλευράς και από τη στιγμή που θα έχουμε την απάντηση της αρμόδιας χώρας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα πρόσφατα γεγονότα. Ευχαριστώ κύριε Μωράης από την Σίλβη Κιγιόμ η κυρία Βίξτρομ. Αλλά δεν τη βλέπω την κυρία Βίξτρομ. Δεν υπάρχει η κυρία Λάμπερτ εδώ, ούτε ο κύριος Κίρκοφ, ούτε ο κυριάκος Τριανταφυλλής. Κύριε Μπρόξ, εσείς τουλάχιστον είσαστε εδώ. Ε, είμαι εδώ. Δεν μιλώ εξ ονόματος των απόντων, λέει ο κύριος Μπρόξ. Μιλάω προσωπικά. αν ήμουν πολίτης οποιασδήποτε από τις χώρες αυτές που αναφέρονται, εγώ θα έθετα το ερώτημα του κατά πόσον εμείς, αυτοί δηλαδή, θα είχαν πραγματικά κάποια ανάγκη για αυτό το γραφείο υποστήριξης του ασύλου, αν έχουν πίεση από ετούντε ασύλου. Γιατί ζητούμε λοιπόν τη συνεργασία τους, απλώς του ζητάμε να δώσουν χρήματα και στέγαση για τους ετούντε ασύλου που <clears throat> έρχονται σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πόσοι Ετούντε άσυλο έχουν έρθει στην Ευρώπη κατευθείαν από τη χώρα από την οποία φεύγουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ε, χερσαία σύνορα με τις χώρες αυτές. Αν περάσουν τις πρώτες ασφαλείς χώρες, μπορεί να ήταν πραγματικοί ετούντε ετούντες ασύλου, αλλά τώρα γίνονται απλώς επιλεκτικοί μετανάστες. Φεύγουν πολλοί από χώρες της Αφρικής που υποφέρουν από τη δημοκρατία που δημιούργησε εκεί, μέσα σε εισαγωγικά, οι, Ευρωπα... οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν περάσει πολλέ χώρε προτού θέσουν τον εαυτό του σε κίνδυνο σε πλοία τα οποία πολλέ φορέ βυθίζονται. Είναι ηρωνικό ότι γίνεται λοιπόν αυτή η συζήτηση μόνο τρει ή τέσσερι μέρε μετά από το ελβετικό δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα τη Κυριακή δεν είχε να κάνει με το άσυλο, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το κλίμα που επεκράτησε εκεί ήταν σαφές. Ευχαριστώ κύριε Μπρόντς. Η Κομισιόν και η Προεδρία εφόσον θέλουν να συμβάλλουν στη συζήτηση, η Κομισιόν, ο κύριος Κατότ, ο Κατότ. Έχετε το λόγο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματα και τα σχόλια που διατυπωθήκαν για αυτή τη συμφωνία, για την πρόταση συμφωνίας με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, την Ορδία και την Ισλανδία για τη συμμετοχή τους στο σύστημα, στο γραφείο για την υποστήριξη του συστήματος ασύλου, όπως είπε και ο εισηγητής, η Κομισιόν τονίζει τη σημασία του να συμμετέχουν και οι συνδεόμενες χώρες, η στο σύστημα αυτό του Δουβλίνου και είναι πολύ θετικό να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστες πρακτικές και άλλες συναφείς ε, ενέργειες, πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης κτλ. Απαντών στο γενικό ερώτημα σε σχέση με το δημοψήφισμα της Ελβετίας. Θα ήθελα να πω εξ της Κομισιόν ότι τα συμπεράσματα αυτού του δημοψηφίσματος είναι υπό εξέταση από την Κομισιόν. Η ελβετική κυβέρνηση τώρα θα πρέπει να εφαρμόσει πλήρως την απόφαση η οποία ελήφθη από τον λαό της Ελβετίας και η Κομισιόν θα ανατάμει με μεγάλη προσοχή οποιαδήποτε απόφαση στην οποία θα καταλήξει η ελβετική κυβέρνηση. Να υπογραμμίσω επίσης ότι υπάρχει μια μνήα, μια πρόνοια σε αυτή τη συμφωνία που έχουμε με την Ελβετία που συνδέει την ε, συμμετοχή στο γραφείο υποστήριξης με την ε, συμμετοχή της ε, Ελβετίας, Λιχτενστάιν και των άλλων χωρών στο σύστημα του Δουβλίνου. Αυτό σημαίνει ότι αν οι χώρες αυτές δεν συμμετέχουν στο σύστημα του Δουβλίνου τότε και η συμφωνία για το γραφείο υποστήριξης και αυτή θα πάψει να ισχύει. Για το θέμα του αν υπάρχει πίεση ετούντων ασύλων στις χώρες αυτές, η Κομισιόν θα ήθελε να υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι χώρες αυτές έχουν επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη συμφωνία Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έρχονται κατευθείαν στις χώρες αυτές και ζητούν άσυλο. Η Νορβηγία, παραγματικά χάρη, έχει υποδεχθεί πρόσφατα πολλούς ε, ετούντες άσυλο από τη Συρία και πιστεύει η Κομισιόν ότι αυτές οι συμφωνίες μπορούν να είναι αμοιβαίας ωφέλειας και για τις δύο πλευρές. Ελπίζω να απάντησα στο ερώτημα των εντύμων μελών του Κοινοβουλίου και μπορώ να επανέλθω αν χρειάζεται. Κοιτάξτε κύριε Κατώτη, εγώ ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Όλοι είχαμε στο μυαλό μας το δημοψήφισμα που έγινε το, την Κυριακή στην Ελβετία ήταν πηχαίοι οι τίτλοι για το αποτέλεσμα αυτού του δημοψήφισματος και δημιούργησε ανησυχίες σε όλους μας οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν στην ευρωπαϊκή διαδικασία, τα ευρωπαϊκά ιδανικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, σημαντικό <clears throat> παίκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα πρέπει να την χάνει σεβασμού από όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις στενές. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποιες είναι οι προοπτικές και ποιες είναι οι νομικές συνέπειες που θεωρεί η Κομισιόν θα προκύψουν από το δημοψήφισμα αυτό. Θέλετε να επεκταθείτε στο σημείο αυτό. Ελπίζω να μπορέσω να διευκρινίσω περαιτέρω τα πράγματα. Νομίζω ότι το σημαντικό στοιχείο που ήδη υπογράμμισα είναι η σχέση με το σύστημα του Δουβλίνου. Δηλαδή, αν η Ελβετία σταματήσει τη συμμετοχή της στο σύστημα του Δουβλίνου, αυτό αυτομάτως θα έχει σαφή συνέπειες για την ε, εφαρμογή αυτής της διευθέτησης, αυτού του συστήματος. Η ανάλυση του δημοψηφίσματος στην Ελβετία σε σχέση με τη συμμετοχή της Ελβετίας σε διάφορες στοιχείες της ε, πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενώσεω είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα σαν αποτίμηση. Είναι κάτι που ξεπερνάει, Η συνέπεια είναι κάτι που ξεπερνάει ε, αυτή τη συζήτηση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιμένει τι θα κάνει η ελβετική κυβέρνηση. Πώς θα εφαρμόσει αυτή την απόφαση. Ακόμα δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση από την ελβετική κυβέρνηση περί εφαρμογής των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος. Άρα δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Περιμένουμε την απόφαση της ελβετικής κυβερνήσεως. Η απόφαση θα αναλυθεί προσεκτικά και για αυτό το θέμα που συζητάμε και για τις ε, σχέσεις σε θέματα εσωτερικών και θα ενημερωθεί η κυβέρνηση για εδήποτε αποτελέσματα της σχετικής αυτής αναλύσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σημειώνουμε, λέει ο Πρόεδρος, τα όσα είπατε. Η Ελληνική Προεδρία, θέλετε να πείτε κάτι, να πάρετε το λόγο. Πάρτε το λόγο, έχει το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την Ελληνική Εκπροσωπεία και ευχαριστούμε ειλικρινά τον εισηγητή για τις εκθέσεις θεωρούμε ότι η ρύθμιση συμμετοχή των συνδεδεμένων ε, μελών ε, ε, στο σύστημα ΕΑΣ είναι χρήσιμη. Σας ενημερώνω δε ότι εχθές το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έλαβε τις σχετικές αποφάσεις για την υπογραφή ω σημεία α. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. τώρα. Η κυρία Μετσόλα, ε, θέλετε να λάβετε το λόγο και πάλι. Για να εξαντλήσουμε το χρόνο που έχουμε προβλέψει για το θέμα αυτό, είναι και τεχνικό. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Το μικρόφωνο τη κυρίας Μετσόλα έκλεισε. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Και έκλεισε το μικρόφωνο τη κυρία Μετσόλα. Δεν ακούγεται καθόλου, δεν υπάρχει μικρόφωνο. Ε, ναι, και εγώ προσβλέπω σε μια ταχεία ολοκλήρωση αυτή τη διαδικασία. Ε, Τούτων λεχθέντων πάντω θα ήθελα πιο πολλέ λεπτομέρειε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν θα έχει ολοκληρώσει την ανάλυση τη σχετική με τι ε, συνέπειε του δημοψηφίσματο τη προηγούμενη Κυριακή και βέβαια, όπω είπε και ο κύριο Μωρέ, από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Προ το παρόν όμω το αφήνουμε εκεί το θέμα. Καλώ λέει ο Πρόεδρος και έχουμε εσείς το χρόνο να προχωρήσουμε στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με την υλοποίηση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση προγράμματος δράσης σε θέματα κατά της ανταλλαγών και συνδρομής για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη. Το λεγόμενο πρόγραμμα Ρίκλης. Το ξέρω. και θα ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή Σκιώδης και Επιτροπή Προεδρία. Πρώτα όμως ο κύριος Δίας Δεμέρα, εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση κανονισμού που μας απασχολεί εδώ έχει σαν στόχο να διευρύνει στα κράτη-μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στο, στη ζώνη του ευρώ την εφαρμογή του προγράμματος Περικλής 2020 για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι απαραίτητες γνώσεις σε χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Δανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχική Δημοκρατία και η Σουηδία σας αναφέρω αυτές τις πληροφορίες και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η περικλήση 2020 είναι η συνέχεια ενός προγράμματος το οποίο είχε δημιουργηθεί από το πρόγραμμα 2001-2003 του Συμβουλίου και όπως ξέρετε είχε στη συνέχεια περάσει από διάφορες τροποποιήσεις με τον βασικό στόχο του να υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα τα οποία αποτελεσματικά αποτελούν μέτρα προστασίας του ευρώ κατά της κυβδηλίας και παραχάραξης. Υπήρξαν σχετικά 7 ή 8 εκθέσεις για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά τη νομική βάση της πρότασης αυτής, βασιζόμαστε στα άρθρα 133 και 139 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ε, εφαρμογή όμως της διεύνησης του προγράμματος Περικλής που θα πρέπει να κάνουμε η πρόταση κανονισμού <clears throat> βασίζεται στο άρθρο 352 της ίδιας αυτής συνθήκης. Οι αξιολογήσεις που έχει κάνει ο ίδιος ο Περικλής <clears throat> το 2004 και το 2011 καταδεικνύουν ότι το πρόγραμμα αυτό επέτυχε τους στόχους του <clears throat> και πρέπει να συνεχιστεί. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι η επέκταση του προγράμματος αυτού στα 10 κράτη-μέλη που αναφέρα <clears throat> προηγουμένως θα επιτρέψει τη βελτίωση αυτού του προγράμματος βοηθώντας και την ενίσχυση της ε, αποτελεσματικότητας του προγράμματος αυτού για την ε, ε, καταστολή της παραχάραξης και κυβδηλίας. Και τέλος, η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος δεν δημιουργεί προβλήματα διότι δεν είναι υψηλή χρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο είναι ασήμαντο αν λάβουμε υπόψη την αποτελεσματικότητα που μπορεί να προκύψει και τις προσπάθειες που καταβάλει η όλα Αυτά θέλω να πω λοιπόν κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δίας μέρα Θα έχουμε λίγο χρόνο για τους σκιώδεις. Κυρία Μάκντάια, έχετε πρώτη το λόγο. Ε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς. Θα γνωρίζετε ότι μιλώ συσυγήτρια για το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος Περικλής. Ευχαριστώ τον κύριο Ντίας Δεμέρα για τη δουλειά που έκανε για το πρόγραμμα Περικλής επίσης. Ήταν άριστη η συνεργασία μας και υποστηρίζω απόλυτα τα όσα μας είπε. Είναι σημαντικότατο το ότι το πρόγραμμα Περικλής επεκτείνεται και στα κράτη-μέλη εκείνα που δεν έχουν το ευρώ σαν νόμισμά τους. Μας επηρεάζει όλους, όλοι ταξιδεύουμε εντός της Ευρώπης. Άρα είναι σημαντικότατο κάθε χώρα να μπορεί να προστατεύει το ευρώ κατά παραχάραξης. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τα κράτη-μέλη που έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Επηρεάζει όλους μας. Είναι σημαντικότατο λοιπόν να επεκταθεί το σύστημα και σε χώρες όπως η δική μου. Επίσης, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Δεμέρα. Πράγματι, είναι πολύ ε, οικονομικό πρόγραμμα, δεν χρειάζεται πολλά χρήματα, χρησιμοποιείται άριστα και είναι η αποτίμηση του προγράμματος, της λειτουργία του είναι θετικότατη μέχρι τώρα. Υποστηρίζω 100% αυτά που προτείνει ο κ. Δεμέρα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κυρία Μάκιντάρ. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Πιερίνη. Κύριε Πιερίνη, κυρία Πιερίνη. Α, όχι, συγγνώμη, ο κύριος Μπρόντς έχει να πει κάτι. Έχετε το λόγο, κύριε Μπρόντς. Ε, μην ανησυχείτε, δεν χρειαστεί να με ξαναδείτε από τον Απρίλιο και μετά γλιτώνετε. Όχι, παρακαλώ, περάστε. Λοιπόν, δεν υπάρχει εμβολία ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με το θέμα του νομίσματος ε, ξεπερνούν ε, βέβαια τα όρια των κρατών που χρησιμοποιούν το νόμισμα αυτό ως κοινό νόμισμα και ως εκ τούτου θα πρέπει να επεκταθεί το πρόγραμμα Περικλής 2020 και στα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Όπως υπόθηκε, 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκτό της Ευρωζώνης, έχουν το εθνικό τους νομισμό η καθεμιά και πρέπει να προστατευθούν από την παραχάραξη και εκείνες όπως και οι χώρες της Ευρωζώνης. Λαμβάνει μέτρα για την προστασία των νομισμάτων, των εθνικών αυτών νομισμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα προστατεύσει από από την παραχάραξη με 7.344.000 για την εφαρμογή του προγράμματος περικλείσε για μια επταετία αν δεν κάνω λάθος στο ποσό λέει ο μιλητής μπορεί να μην είναι πολλά ποσά μπορεί όπως λέει ο κύριος Δίας Δεμέρα να είναι μηδαμινά τα ποσά αλλά εάν μπορεί να αυξήσει το ποσό αυτό κατά 10% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με καταξιδότηση πράξη θα πρέπει να λάβει υπόψη και το γεγονό ότι το χρηματοδοτεί ο προπολογισμό όλων των κρατών που συμβάλλουν σε αυτόν και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μεγαλύτερη συμβολή. Άρα θα πρέπει και για την προστασία όλων και το συμφέρον όλων να προστατευτούν όλα τα εθνικά νομίσματα, όχι μόνο το ευρώ και άρα ίσως ιδιαίτερα οι χορηγοί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που δεν θα πρέπει μόνο να πληρώνουν αλλά να έχουν και προστασία για το εθνικό τους νόμισμα. Για τα δέκα άλλα νομίσματα. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα λύσει η Επιτροπή. Κύριε Πιερίνη, θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Και το όντι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμέρα και την κυρία Μάκιντάιρ για την ε, υποστήριξή τους και για τη συμβολή βέβαια τον κύριο Μπρόνς η επέκταση σε χώρες εκτός Ευρωζώνης, της προστασίας ε, του ευρώ κατά της παραχάραξης, είναι ένα μέτρο που κατευθύνεται προς την ομοιογενή προστασία ενός νομίσματος κατά εγκληματιών που το επιβουλεύονται. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι η συνθήκη της Γενέβης υποχρεώνει την κάθε χώρα να προστατεύει κάθε νόμισμα, οικείο και ξένο, από κάθε επίθεση ανεξαρτήτως ε, του ποιο νόμισμα είναι αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν ε, αποτελεί εξαίρεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα μέσα που διαθέτει το πρόγραμμα Περικλής ε, αυτά τα χρόνια έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια για να προστατεύσει κάθε νόμισμα, όλα τα νομίσματα με προτεραιότητα ασφαλώς το ευρώ, αλλά καταρτίζουμε όλο το προσωπικό, τους υπαλλήλους που έχουν ε, ασχοληθεί με την αντιμετώπιση παραχάρησης και της κυβδηλίας και βέβαια μαζί με όλες τις χώρες που καταπολεμούν την παραχάραξη, καταπολεμούμε την παραχάραξη κάθε νομίσματος και όχι μόνο του ευρώ. Αυτό πρέπει να το πω με απόλυτη σαφήνεια. Καταρτίζουμε λοιπόν ειδικού ε, αξιωματούχους για την καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ, έμεσα όμως τους καταρτίζουμε και στην καταπολέμηση της παραχάραξης εθνικών νομισμάτων. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Βέβαια η οδηγία για την προσοχή του ευρώ στόχο έχει να προστατεύσει κάθε νόμισμα κατά της παραχάραξης. Τούτου λεχθέντος. Ευχαριστώ την Επιτροπή στο σύνολό της για την μεγάλη προσπάθεια και την αντίληψη, την ε, αποδοχή της ανάγκης να προστατευθεί το ευρώ κατά της παραχάραξης. Ελπίζουμε και εμείς να προχωρήσει σε ταχύτατη έγκριση η πρόταση και βέβαια σε κύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών όπου αυτό προβλέπεται. ένα Βασίλειο Φεριπίν και Γερμανία. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να εξασφαλιστεί ομοιογενής προστασία του ευρώ κατά της παραχάραξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πιερίνη, η Ελληνική Προεδρία λαμβάνει το λόγο. Όχι, δεν έχετε σχόλιο. Και ίσως, αν θέλετε κύριε Δίας Δεμέρα να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μακιντάερ για τα θερμά της λόγια και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο της γιατί εγώ συνεργαστεί μαζί της σε άλλες εκθέσεις που έχουν ακριβώς σαν αντικείμενο το θέμα της, προ... της προστασίας του ευρώ από παραχάραξη και εκτιμώ και τα σχόλια του κυρίου Μπροντ. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό το οποίο είπα σε σχέση με τον εκπρόσωπο της ΟΛΑΦ. Πρόκειται, τονίζω και πάλι πρόκειται για μια προστασία που αφορά όλα τα ευρωπαϊκά νομίσματα, αλλά ο Περικλής, το πρόγραμμα Περικλής αφορά μονάχα στην προστασία του ευρώ. Κύριε Μπρόνς, αναλαμβάνω την πρόκληση αν θέλετε να κάνετε μια νομοθετική πρωτοβουλία και προτείνεται ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την προστασία της αλβιονικής λύρας, εγώ θα το υποστηρίξω χωρίς καμία αμφιβολία, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νόμισμα. Γιατί είναι όλα αυτά, πω και το εξή. Υποστηρίζω ιδιαίτερα και εκτιμώ το επαγγελματικό έργο που έχει κάνει η ΟΛΑΦ σε σχέση με τα θέματα αυτά στην προσπάθειά της και στο ζήλο της για να, προσπαθεί, το νόμισμα των 18 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανώνει ο ΛΑΦ κύκλους κατάρτισης προς το, την κατεύθυνση διαφόρων ε, υπαλλήλων και φορέων και αυτών που ασχολούνται που ασχολούνται με την προστασία του ευρώ από κυβδηλία. Και αυτό γίνεται σε πολύ ευαίσθητα μέρη στον κόσμο. Χαίρομαι λοιπόν που με προσκαλούν να είμαι μαζί τους. Χάρη στις ε, συνεργασίες που έχουμε κάνει σε νομοθετικό επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να είμαι μαζί σας και πέραν του Ματίου συνεργαζόμενος με την ΟΛΑΦ στην Λατινική Αμερική. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δία σήμερα. Περνάμε στο επόμενο σημείο λοιπόν. Το επόμενο σημείο είναι το 16. Έχουμε μια μελέτη μπροστά μας του Τμήματος Διαμόρφωσης Πολιτικής ανάπτυξη χώρου ποινική δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσουμε την παρουσίαση από τη δόκτωρα Μαριάν Βουίτ, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Δικαστικής Δίκησης στο Birmingham, στη νομική σχολή του Μπέρμιγχαμ, και τη δόκτωρα Μέχτιλτ Μπάουμαν. Η δόκτωρα Μέχτιλτ Μπάουμαν λοιπόν θα αναφερθεί στο θέμα αυτό. Έχουμε την ε, έκθεση, παραδόθηκε η μελέτη μάλλον και μοιράστηκε στα μέλη το ποινικό δίκαιο. Είναι πολύ ευαίσθητος νέος νομικός τομέας. Αναφέρεται στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσης, συνθήκη της Είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα προόδου στην ευρωπαϊκή ιστορία τελευταία τέσσερα χρόνια εγκρίναμε διάφορα μέσα ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση σε, ε, σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών, εμπορίου παιδιών, διάφορες οδηγίες, το ευρωπαϊκό ένταλμα, οδικό χάρτη για τα διάφορα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες για προσφυγή στη δικαιοσύνη και η δημιουργία χώρου ποινική δικαιοσύνης δεν έχει ολοκληρωθεί, ε, τώρα ξεκίνησε, εκρεμεί Ακόμα η πρόταση για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία, σημαντικότατο θέμα και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καλύπτεται αυτό. Πληροφορίες χρειάζονται για την ένωμη τάξη των διαφόρων κρατών μελών όσον αφορά την ανάπτυξη αυτού του νεογέννητου τομέα α, χώρου, ενίου χώρου ποινική δικαιοσύνης. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτή η μελέτη της δόκτωρος Μαρίαν Βέιτ και της δόκτωρος Μακτίλτ Μπάουμεν που θα ακούσουμε ότι αυτή η μελέτη θα τονίσει τη σημασία του θέματος. Σας ακούσουμε λοιπόν τι έχουν να μας πούνε. κυρία Βέιτ καταρχάς, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που ανέθεσε αυτή τη μελέτη ε, και ενδιαφέρθηκε για την άποψη των πανεπιστημιακών για το θέμα. Είμαι η Μαριάν Βέιντ, είμαι από το Πανεπιστήμιο του Birmingham ε, όπως παρουσιάστηκε από την νομική σχολή και έγινε η μελέτη μαζί με το αντίστοιχο Ινστιτούτο του Βερολίνου υπό την ηγεσία της δόκτωρος Μπάμον που είναι παρούσα και ευχαριστώ και πολλούς άλλους ακαδημαϊκούς ε, που οι μελέτες τους και το έργο τους μας επέτρεψε να ετοιμάσουμε τόσο γρήγορα αυτή τη μελέτη και ευχαριστούμε και τους βοηθούς ε, μία από τους βοηθούς είναι εδώ παρούσα ξέρω ότι υπάρχει χρονική πίεση θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα βασικά σημεία και τις βασικές απειλές που ενατόπισα. Έχετε αντίγραφο της μελέτης όλοι σας και μπορείτε να τα εξετάσετε με την ησυχία σας. Δυστυχώς υπήρξε πρόβλημα το μικρόφωνο αλλά επεκαταστάθη. Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να τονίσω είναι ότι υπάρχει ένα βασικό θέμα που τίθεται στην κατάσταση που δημιουργείται μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ανώσεως Στη στήκη της Αβώνας βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να επιβάλλουν κάποια όρια όσον αφορά το εύρος του, ευρωπαϊκού, ε, του χώρου του ευρωπαϊκού για την ποινική δικαιοσύνη. Και όπως αναφέρεται και στην ανάθεση της μελέτης και στις ιδέες που δώσαμε τη μελέτη, εστιαστήκαμε όχι μόνο στα εγκλήματα που ήδη καταγράφονται, αλλά και ποιο είναι το νόημα τη φράση που έχω τονίσει. Ποια είναι τα ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, εγκλήματα με δυσυνοριακό χαρακτήρα. Άρα υπάρχουν όρια όσον αφορά την εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ενώσης στην ποινική δικαιοσύνη. Πρέπει να καθοριστούν τα όρια για τη λειτουργία τη επιτροπή ΛΥΜΠΕ εντό του Κοινοβουλίου και στην νομική διαδικασία. Το να μπορεί να πει κατά πόσο είναι εκτό ορίων, εκτό ορίων κάποιο αδίκημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω λοιπόν να βλέπετε διαφάνεια. Καλώς. Καταρχάς, βλέπουμε τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Αυτή η ιδέα των σοβαρών αδικημάτων, ε, τι νόημα, αν έχει νομικό νόημα. Πριν ξεκινήσουμε τη μελέτη που υποβάλαμε, είδαμε ότι δυστυχώς σοβαρά αδικήματα είναι σημαντική φράση από πολιτική σκοπιά, αλλά δεν νομικός όρος που βοηθάει που πουδενή να καθορίσουμε την έννοια του σοβαρού και μη σοβαρού αδικήματος. Βασικό πόρισμα της μελέτης σχετικά με αυτό είναι το εξής. Αν δείτε τις ε, ποινικέ δικαιοδοσίες στα την ποινική νομολογία στα κράτη μέλη, βλέπει κανείς ότι σοβαρά αδικήματα είτε έχουν καθοριστεί για ειδική αντιμετώπιση κάποιες μορφές σοβαρών αδικημάτων, κυρίως τρομοκρατικές πράξεις, οργανωμένο έγκλημα, έχουν απομονωθεί για συγκεκριμένη αντιμετώπιση ή θα δείτε ότι η νομολογία έχει ε, προσαρμοστεί στα λιγότερα σοβαρά αδικήματα, ώστε ο χρόνος των δικαστηρίων και οι αναλυτικές εξυχνιάσεις να αφιερώνονται των εγκλημάτων να αφιερώνονται στα σοβαρά εγκλήματα. Άρα βλέπουμε αρνητικό ορισμό και δυστυχώς τίποτα που να μπορεί να μας οδηγήσει να πούμε θετικό τρόπο ότι αυτή είναι μια ευρωπαϊκή έννοια του σοβαρού εγκλήματος. Στις διαφάνειες δείχνω τους δείκτες περίπου όσον αφορά το θέμα του σοβαρού εγκλήματος. Λέμε λοιπόν υπάρχουν αδικήματα και εγκλήματα για τα οποία τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα προβληματικά για το ποινικό δίκαιο και τι ποινικέ έρευνε και αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο. Όποιο ασχολείται με θέματα ποινική δικαιοσύνη θα εκπλήσεται βλέποντα ότι είναι οι πιο αόριστε έννοιε ε, της τρομοκρατίας και του πολύ σοβαρού αδικήματος. Έχουμε ειδικέ διαδικασίες του σοβαρού αδίκημα, όχι δεν έχουμε. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ειδικέ ιδιωτότητες όπως να μπορεί κανείς να τοποθετηθεί όσον αφορά το αδίκημα και να γίνουν κάποιες διαπραγματεύσεις για την τελική ε, απόφαση. Αλλά δεν μπορούμε να καθορίσουμε ποια αδικήματα θεωρούν ως μη ιδιαίτερα σοβαρά τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν έχουμε θετική ε, αντιμετώπιση για να μπορούμε να το καθορίσουμε με βάση το άρθρο 83 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λοιπόν, σε περιπτώσει τρομοκρατία και οργανωμένου εγκλήματο, κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι ύποπτοι για τέτοια αδικήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, χάνουν κάποια δικαιώματά του όσον αφορά τη δικαιοσύνη και είναι πολύ συντηρητικά κάποια κράτη-μέλη σε αυτή την αντιμετώπιση. Σοβαρό αδίκημα, σοβαρό έγκλημα στι περισσότερε περιπτώσει δεν οδηγεί σε απώλεια δικαιωμάτων ή χαλαρή αντιμετώπιση, πιο χαλαρή εφαρμογή των βασικών αρχών του συστήματος ε, του νομικού και της ποινική δικαιοσύνης. Λοιπόν, το πρώτο πόρισμα ποιο είναι, ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει καθαρό ορισμό, αυτόνομο ορισμό, τι είναι το σοβαρό έγκλημα και ποια είναι τα νόμιμα όρια όσον αφορά του ευρωπαϊκού συστήματος, του χώρου του ευρωπαϊκού για το ποινικό δίκαιο. Έχουμε αρκετές ενδείξεις στον αφορά αυτά τα όρια. Ήδη συζητήσαμε. Ζωηρότατη συζήτηση έγινε μεταξύ κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε δύο πράγματα. Έχουμε ευρωπαϊκή ποινική δικαιοσύνη, δηλαδή ουσιαστικό δίκαιο, αλλά και θεσμικά μέτρα, διαδικαστικά μέτρα που κινούνται σε δύο άξονες. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κυβέρνησης που ρυθμίζει συμπεριφορές όπως τα ξέρετε, όσον αφορά το περιβαλλοντικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε ότι καμιά φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν, σαν επίπεδο διακυβερνητικό ρυθμίζει συμπεριφορές. Άρα χρειάζεται ένα εργαλείο, το ποινικό δίκαιο. Υπάρχουν κάποιοι τομείς πολιτικής που είναι στις δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που ίσως να χρειάζονται διευθέτηση μέσω ποινικού δικαίου. Και χρειάστηκε ποινικό δίκαιο για την προστασία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να προστατεύονται τα συμφέροντα και αξίες της. Κυρίω ανθρωπολογικώ οι κοινέτητε χρησιμοποιούν την ποινική δικαιοσύνη για να προστατεύουν και να υπερασπίζονται τι πιο βασικέ αρχέ. Άρα, πρέπει να σκεφτούμε ποιε είναι αυτέ οι βασικέ αρχέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συζητήσει που διεξάγονται για τι προτάσει για το χώρο του ποινικού δικαίου εξετάζουμε τα οικονομικά συμφέροντα. Λοιπόν, όσο με αφορά, αυτό είναι ένα από τα έμβρια, τα δίδυμα έμβρια που βρίσκονται στο άρθρο 86 Συνθήκη τη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Στο άρθρο 86 τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ενώσεω αναγνωρίζεται ότι τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο μπορούν να επεκτείνουν την, ε, το χώρο αυτού του χώρου ποινική δικαιοσύνη. Αναγνωρίζεται την τελευταία 15 ετία η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εξειδικευτεί ω ιδιαίτερο όσον αφορά την απόδοση σε υπερεθνικό επίπεδο τη δικαιοσύνη. Πώ το βλέπω αυτό θεωρητικά. Οι τέσσερι ελευθερίε που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώ μπορεί καμιά φορά να θεωρηθούν σαν παράγοντε διευκόλυνση παρανόμων δραστηριοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν διατείνομαι ότι οι τέσσερι ελευθερίε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω αντιπροσωπεύουν τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και εκείνε που η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να υπερασπιστεί σαν δικέ της πολύ βασικές αρχές βάσει με την επιφύλαξη αρχής επικουρικότητας και σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Μπορούμε τώρα μετά τη Λισαβόνα να θεωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι επίπεδο διακυβέρνησης που έχει ηθικές ευθύνες έναντι των πολιτών. Και θα επανέλθω σε αυτή την ιδέα τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε επίπεδο διακυβέρνηση και των πολιτών που είναι αποδέκτε σε άμεση σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είναι κάτι σημαντικό κατά την άποψή μου όσον αφορά την απόδοση τη δικαιοσύνη στον ποινικό τομέα. Δηλαδή βρήκα, είμαστε στη φάση που μπορούμε να μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ένα επίπεδο διακυβέρνησης με ηθικές ευθύνες. Για λόγους ρεαλιστικούς και πολιτικούς βέβαια, το καταλαβαίνω ότι δεν εστιάζεται επ' αυτού η συζήτηση τώρα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται επί των οικονομικών συμφερόντων. Αυτό είναι κατανοητό. Όπω τα βλέπω εγώ τα πράγματα, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι εδήποτε χώρο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για το ποινικό δίκαιο έχει επιπτώσεις σε συνταγματικό επίπεδο για τους δικαιούχους συνταγματικών δικαιωμάτων. Να σας δείξω ποιο είναι το εύρος κάλυψης της μελέτης αυτής, να αναφερθώ στο εξή. Η μελέτη έχει συγκριτική βάση και θέλαμε να εμπνευστούμε για κανόνες και κανονισμούς από τα κράτη-μέλη για να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θεμελιώδες όμως πόρισμα είναι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και επικοινομορφία, πολλές διαφορές μεταξύ κρατών μελών και αναφέρω παραδείγματα. Λοιπόν. Έχω τέσσερις διαφάνειες πιστεύω θα σας δείξουν ποια κεντρική σημασία έχουν τα δικαιώματα της περάσπισης. Δεν ε, πιστεύω ότι θα προλάβετε να τα δείτε όλα, αλλά στα σημεία 1 έως 1, 5 και μετά στην έκθεσή μας μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά. Ε, αν δείτε λοιπόν ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία θεωρούν ε, κεντρική σημασία στα κράτη-μέλη, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο φάσμα. Έχουμε το δικαίωμα ε, το, έχουμε το τεκμήριο της το δικαίωμα να, να πει κανείς ψέματα για να προσπαθήσει τον αυτό του, την αξιοπρέπεια του ατόμου, κεντρική σημασία σε ορισμένε συνταγματικές τάξεις, το δικαίωμα για ε, υπεράσπιση, την ισότητα των όπλων στην ε, δίκη και μια, μια σειρά από άλλες ε, αρχές. Ακόμα λοιπόν και όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποια είναι η ουσία, ποιος είναι ο πιο σημαντικός τομέας, η ομάδα δικαιωμάτων ε, για την υπεράσπιση ε, είναι δύσκολο να το, να το πείσουμε ένα κοινό. Επομένω, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την ε, διαδικασία τα δικονομικά, στα δικαιονομικά δικαιώματα, την ισότιμη υπεράσπιση, αλλά και πολλά άλλα που θεωρούνται ιερά από ενώμες τάξεις. Μας έφυγε λίγο η διαφάνεια. Για να επιδείξω ακόμη περισσότερο τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, βλέπετε στην έκθεση στο 9, σελίδα 34, και παράδειγμα του καταμερισμού ή του επιμερισμού καλύτερα αρμοδιότητων μεταξύ ε, δικαστηρίου, ε, ανακριτικής αρχής και ανεξάρτητης δράσης αστυνομία δικονομικά. Δηλαδή, ποιος έχει πιο κομμάτι αρμοδιότητας για την διαχείριση των δικαιωμάτων ή την ε, εποπτεία της στήριξης των δικαιωμάτων, που πάλι παρουσιάζει πολύ μεγάλη ποικιλία, όπως τον αναμενόμενο. Αν μπορούσαμε να πάμε πίσω... Η τεχνολογία μας έχει καταλήψει από ό,τι φαίνεται. Ένα από τα κεντρική σημασία δικαιώματα, πώς το εντοπίζουμε εμείς ως πολύ σημαντικό, είναι ότι στα συστήματα της ποινική δικαιοσύνης που έχουν αναπτυχθεί του τελευταίους τέσσερις αιώνε για ορισμένες δικαιοδοσίες ε, έχουν αναπτυχθεί σε διάλογο μεταξύ ηγεμόνα και υπηκών και έτσι έχει προκύψει μια μορφή κοινωνικού συμβολέου με προσδοκίες από πλευράς του πολίτη λόγω των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει ή που του έχουν χορηγηθεί. Ένα λοιπόν από τα ζητήματα και η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το δικαίωμα της ε, υπεράσπισης να συμμετέχει ενεργά στις ε, ανακριτικές έρευνες και αυτό το έχω μέσα στο κείμενό μου. Τη διαφάνεια τώρα δεν μπορούμε να τη βρούμε εύκολα, αλλά πάντως 50% των κρατών μελών θεωρούν ότι το άτομο, ο πολίτης, ο ιδιώτης που εμπλέκεται σε μια ποινική διαδικασία, πιστεύει και θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει ενεργά στην ανάκριση όχι όμως μόνο ο κατηγορούμενος, αλλά και, για να περάσω τη διαφάνεια με τα θύματα, και τα θύματα έχουν ε, δικαιώματα και σε ορισμένες περιπτώσεις και δικαίωμα συμμετοχή στην ανακριτική διαδικασία. Βλέπετε εδώ τα δικαιώματα της υπεράσπισης για συνδρομή στην ανακριτική διαδικασία. Αλλά αν δείτε και πώς ένα σύστημα δικαιοδοτικό εξυπηρετεί τον πολίτη, τη τελευταία μία-δύο δεκαετίες έχουν εγερθεί και διεκδικήσεις για συμμετοχή των θυμάτων, είτε πρόκειται για το ενδοτικό δίκαιο, είτε πρόκειται για το αναγκαστικό, στην διερεύνηση μιας υπόθεσης. Και εδώ πάλι έχουμε τεράστιες αποκλήσεις μεταξύ κρατών μελών για το πώς βλέπουν και πώς υλοποιούν αυτά τα δικαιώματα και τις εκδικήσεις. Επίσης, πολύ σημαντικό, μέγιστος αποδεκτός χρόνος φυλάκισης, όπου πάλι βλέπουμε διαφορές στα κράτη-μέλη. Βέβαια, η ε, επιμέτρηση της ποινής έχει πολύ μεγάλη σημασία, εν προκειμένου. Και για να κοιτάξουμε ε, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει, να αναλάβει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ποινικού δικαίου με τόσο μεγάλη ποικιλία διαφορετικών λύσεων στις ένωμες τάξεις, υπάρχει κίνδυνος, από ό,τι διαπιστώνουμε, να θεωρηθεί ότι μειώνονται οι προδιαγραφές σε σχέση με αυτά τα οποία περιμένουν οι πολίτες, εάν επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κάποια λύση. Η προφανή λύση βεβαίω είναι να πει κανεί ότι ο χώρο τη ποινική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τι ύψιστε δυνατέ προδιαγραφέ. Ξέρω ότι αυτό στι συζητήσει μεταξύ κυβερνήσεων μπορεί να φαίνεται ω έργο Ηράκλειο, αλλά μπορεί και να μας εμπνεύσουν διαφορετικά συστήματα, γιατί βλέπουμε ότι το FBI και γενικά τα κεντρικά συστήματα δικαιοδοσίας έχουν ενισχύσει το, την προστασία ε, των δικαιωμάτων των πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επί παραδείγματι, η επίκληση της, ε, του, της διατάξεως, τέλος πάντων της αρχής ε, που προκύπτει από την ομολογία Μιράντα, έχει βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου σε επίπεδο ομοσπονδιακό, όπου γίνεται επίκληση στα δικαστήρια. Επίσης, όταν μιλάμε για την δουλειά της ε, ποινική δικαιοσύνης και πόσο ε, ευαίσθητη είναι αυτή, πόσο μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα των πολιτών, δεν μπορούμε να λησμονήσουμε όλα τα θέματα που προκύπτουν από τις συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Η προσωρινή κράτηση ε, πολιτών με διαφορετικούς χρόνους ανακράτος μέλος είναι απαράδεκτη. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται επί παραβιάση των, ε, υποχρεώσεων τους δυνάμει της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στην υπόθεση Άντρου Σίμουνς έχουμε μια σύλληψη και προσωρινή κράτηση σε απαράδεκτες συνθήκες φυλάκισης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μια περίπτωση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ε, επικίνδυνες εξελίξεις για το ευρωπαϊκό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, γιατί αυτό θα αφήσει όμοιρο την ευρωπαϊκή ποινική δικαιοσύνη στα χέρια εκείνων, οι οποίοι θα θέλουν να την κατηγορήσουν για πάνδυνο και θα επικαλούνται ότι είναι πολύ κακές οι προδιαγραφές και η προστασία των δικαιωμάτων. Επίσης, το δικαίωμα για πρόσβαση συνήγορο, όταν ε, για δεκαετίες ακόμη και αιώνες θεωρεί ένας πολίτης δεδομένο το ότι η περίπτωση να βρεθεί ενώπιον του νόμου κατηγορούμενο συνεπάγεται αυτόματα και τη δωρεάν παροχή δικηγόρου από το νομικό σύστημα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να, από το οποίο είναι πολύ δύσκολο να παραιτηθούν οι πολίτες. Δεν μπορείτε να το γνωρίσετε αυτό. Η ε, συνδρομή λοιπόν, η συνδρομή δικηγόρου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα το δούμε και αργότερα. Είναι βέβαιο ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ε, δικαίωμα πάντως, το, το δείχνει και η μελέτη. Η αντιμετώπιση των ανηλίκων έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ευαίσθητο θέμα. Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα τη μεγάλη απόκληση που επικρατεί μεταξύ κρατών μελών για την ε, ποινική ενηλικίωση, για το πότε υπάρχει δηλαδή η ε, δυνατότητα να κατηγορηθεί κανείς για ποινικό αδίκημα 9 ετών πολύ ασύνηθες, 10 ετών ή 16 μετά η ε, ενηλικίωση και η δυνατότητα καταλογισμού, ανάλογα με το κράτος μέλους. Έχουμε μελέτες επίσης για τα ενισχυμένα δικονομικά δικαιώματα. Έχω κάνει την ανάλυση εδώ και το κύριο συμπέρασμα νομίζω της μελέτης είναι ότι η ιδέα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας ή μετάγγιση δηλαδή της ε, συνθήκης στη φάση μετά τη Λισαβόνα θα περάσει μέσα από την ποινική δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς θα πρέπει να επιβληθεί και κάποιο όριο στις ποινικές δικαιοδοσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να επεκτείνεται κατ' ουσίαν σε κάθε αδίκημα η ποινική δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει κάποια αρχή επικουρικότητας και αναλογικότητας. Η εμπλοκή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσδοριστεί με επαρκείς όρους στην ουσία της, αλλά αυτή η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη και σε αυτό το σημείο. Διότι αν θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα επίπεδο διακυβέρνησης με άμεσο σύνδεσμο με τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και σε θέματα ε, πολύ ευαίσθητα και συνταγματικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν συμπέρασμα απευθεία προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Ποινική Δικαιοσύνη έχει λίγο πολύ μέχρι τώρα συνδεθεί με τις εκτελεστικές πράξεις και τα, ε, έχει μετατραπεί σε μια εκτελεστική πράξη και τα κράτη-μέλη την αξιοποιούν για να προωθήσουν δικά τους συμφέροντα. Δεν υπάρχει σύστημα όμως ποινικό σε κράτος μέλος το οποίο να επιτρέπει την ανεξέλεγκτη λειτουργία του εκτελεστικού με κάποιο τρόπο υπάρχει έλεγχο και συνήθω μέσω κοινοβουλίου και γι' αυτό με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε να μιλήσω σε κοινοβουλευτικό χώρο ανταλλαγών το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ευαίσθητε διαδικασίε, συνταγματικά λεπτέ ισορροπίε και δεν είναι δυνατόν να επικρατούν μόνο τα κατασταλτικά, οι κατασταλτικέ επιλογέ των κυβερνήσεων όπω συμβαίνει μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν να χαράξουν μια γραμμή για το πού εμπλέκεται, μέχρι πού εμπαραίτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ποινική δικαιοσύνη και πού σταματάει για να υπάρχει σωστή ισορροπία. Μπορούμε μερικέ φορέ να πούμε ότι θα περιορίζεται στην διευκόλυνση τη συνεργασία μεταξύ των κρατών η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω συμβαίνει μέχρι τώρα, αλλά επίση και σε επίπεδο διακυβέρνηση που θα υπηρετεί τον πολίτη, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναλάβει την ευθύνη για πολιτικέ όπου μπορεί, αλλά και οφείλει να αναγνωρίσει πω πρέπει έχει καθήκον να αναλάβει δραστηριότητες στο επίπεδο της ποινική δικαιοσύνης να προστατεύσει τα θύματα και θα ήθελα να εξεταστεί το κατά πόσον θεωρείται νομικά διαφορετική η ποινική δικαιοσύνη, ε, δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εθνική, διότι εμπλέκει περισσότερα κράτη-μέλη και άρα μπορεί να έχει ε, ένα διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πια πώς θα προστατεύονται τα δικαιώματα των ε, ιδιωτών, πώς θα απονέμεται η δικαιοσύνη και ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, όπως είπα, μας ενδιαφέρει το ζήτημα του κατηγορουμένου, αλλά δεν μπορούμε να λησμονούμε και τα δικαιώματα των θυμάτων. Εάν ο χώρος της ποινική δικαιοσύνης Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθήσει να συνδέεται με την ταχεία απονομή της κατασταλτικής ε, ποινική δικαιοσύνης που μόνο στρέφεται κατά ενός πολίτη, τότε κινδυνεύουμε να δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κατάχρησης ε, θύμα καταχρηστικών επικρίσεων, σκληρών επικρίσεων χωρίς νόημα και αυτό θα ήταν λάθο. Θα πρέπει να μπορεί βεβαίω να διευκολύνει τα κατασταλτικά μέτρα ει βάρο των πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα προστατεύοντα και το πολίτη. Διαφορετικά θα εκτίθεται σε αυτέ τι ε, επικρίσει από κόμματα όπω το UKIP στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματι. Τα κράτη-μέλη δεν είναι το μόνο ακροατήριο για τη λογοδοσία και τη νομιμοποίηση τη δημοκρατική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώ. Ε, υπογραμμίζω με επιφάσιο το γεγονό ότι η σχέση που έχει ο πολίτη ω δικαιούχος κάποιων δικαιωμάτων και συνταγματικών δικαιωμάτων είναι πολύ πιο έντονη μετά τη Λισαβόνα και επειδή αυτές οι διαδικασίες νομικά έχουν διαφορές θα ήθελα να προτείνω παρότι είναι πολύ χρήσιμη και ίσως μπορεί να αποτελέσει και πηγή έμπνευση η σύγκριση διαφορετικών ενόμων τάξεων πρέπει να είναι έτοιμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο μετά τη Λισαβόνα και να αναγνωρίσει ότι υπάρχει δυνατότητα να αναζητήσει και να σχηματίσει αυτόνομα κάποιες έννοιες για το πώς θα εντάξει τον πολίτη στο επίκεντρο του χώρου της ποινική δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε. Δόκτωρ Ρέσα Βέιτ για την εξαντλητική σας παρουσίαση και τόσο ενδιαφέρουσα. Δόκτωρ Μπέρμαν, θέλετε να προσθέσετε κάτι, θέλετε να κάνετε κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις ή όχι. Εάν όχι, Έχει παρουσιαστεί λοιπόν η μελέτη για την ανάπτυξη της ε, ποινική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι θα, θα ήθελαν να λάβουν. Κύριε Μπρόντς, έχετε τον λόγο. Ξέρω ότι θα σας λείψω μετά τον Απρίλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σαφήνεια και την πληρότητα των εξηγήσεών σα, Δεν βλέπω τα πράγματα από την ίδια οπτική γωνία όπως και εσείς. Είμαι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως εναντίον του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως. Συμφωνείτε όμως ότι όσο υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης θα πρέπει η χώρα η οποία εκτελεί ένα τέτοιο ένταλμα θα μπορεί να αρνηθεί να το, εκτελέσει, να το εκτελέσει για λόγους ανεπαρκών στοιχείων, κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Εγώ φυσιολογικά δεν θα υποστήριζα το, την προτινόμενη <clears throat> εντολή έρευνας. Αλλά όσο υπάρχει το ένταλμα αυτό, το θέμα μιας ευρωπαϊκής ε, εντολής έρευνας θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι μειώνεται η δυνατότητα να εκδίδονται εντάλματα ε, έρευνας στις πιο ασθενείς νομικά οι επιπτώσεις, περιπτώσεις. Είναι σωστό αυτό. Υπάρχουν άλλα σχόλια, κυρία Μάκιντα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την δόκτωρα Wade για την θαυμάσια παρουσίασή της. Είμαι μεροληπτική γιατί ήμουν την προηγούμενη Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο του Birmingham μαθαίνοντας πόσο καλά λειτουργεί αυτό το πανεπιστήμιο. Είναι πολύ καλά λοιπόν που έχουμε αυτή τη θαυμάσια παρουσίαση από την νομική σχολή του Βέρμιγχαμ. Όλα αυτά καταδεικνύουν την τεράστια πολυμορφία που υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας βοηθάει ιδιαίτερα να έχουμε όλες αυτές τις διαφορές οι οποίες αναλύονται και παρουσιάζονται με τέτοια σαφήνεια. Ένας από τους χώρους που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι τα θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών. Το θέμα της ηλικία στην οποία γίνονται ε, έχουν την δυνατότητα να κάνουν κάποιες δικαιοπραξίες και την ηλικία των παιδιών τα οποία εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες. αυτό είναι ένας τομέας που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και εκεί θα ήθελα να ξέρω περισσότερο για τις διαφορές που ισχύουν στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι σε τελική ανάλυση η επικουρικότητα θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις μας για το τι ακριβώς είναι εφικτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποια πρέπει να είναι τα δικαιώματα σε επίπεδο κρατών μελών και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε περαιτέρω. Νομίζω ότι η συνεργασία είναι κάτι το εξαίρετο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο συχνά αναγνωρίζοντας πάντα τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη-μέλη και τα προβλήματα επικορικότητας τα οποία από τη δική μου πλευρά είναι πολύ μεγάλη σημασία και το έγγραφο αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να ε, προωθήσουμε τις συζητήσεις μας και ευχαριστώ πολύ την δόκτωρα Wade. Άλλα σχόλια? Εάν όχι, δεν θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Και εγώ να πω κάτι για τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση των ε, αρμοδίων του τομέα. Συζητούμε το θέμα αυτό εκτεταμένα το, ποινικό, το χώρο ποινικού δικαίου, πώς θα συνεργάζεται ο δικαστικός τομέας και όλοι όσοι εργάζονται στον τομέα, αλλά δεν έχουμε τονίσει επαρκώς τη σημασία το να ε, συμμετάσχουν οι ε, επαγγελματίες του τομέα στο όλο σύστημα επαρκώς. Οι, οι νομικοί, οι δικηγόροι, όσοι κινούνται στον τομέα αυτόν. Διότι αν δεν είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα, ούτως ώστε ο νεογέννητος αυτός χώρος ποινικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να είναι αποτελεσματικός δεν θα υπάρχει νόημα όσον αφορά την προσπάθεια. Θέλω τα σχόλιά σας όσον αφορά αυτό το θέμα. Κάθε φορά αναφέρομαι σε αυτό που έχω την ευκαιρία. Έχετε το λόγο, κυρία Βέιτ. Ευχαριστώ εκ νέου. Σας ευχαριστώ για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά σας. Όσον αφορά το πρώτο σχόλιο, βέβαια καταλαβαίνω ότι υπάρχουν διαφορές, σε στις απόψεις όσον αφορά το θέμα. Το βασικό πρόβλημα με το Ευρωπαϊκό Έντομα Σύλληψης ποιο είναι. Πού, ε, πού βρίσκονται ευθύνε όταν την απόφαση για την παράδοση και μετακίνηση του υπόπτου στη δικαιοδοσία στην οποία αισθάνεται πιο άνετα ο κατηγορούμενος σε σχέση με αυτή στην οποία αισθάνεται πιο ευάλωτος. Άρα είναι προς του κατηγορουμένου να θέλουν να συνδυάζονται οι δύο αυτές ακροάσεις. Είναι θέμα πολιτικής προτεραιότητας που τίθεται από το Ευρωπαϊκό Έντομα Σύλληψης. Δηλαδή εμπιστεύεται κανείς την κρίση του συναδέλφου σε άλλο κάτω μέλος. Εγώ δεν είμαι πεισμένη. Ιδιαίτερα βλέπω ποια είναι η εμπειρία όσον αφορά ε, όσον αφορά το θέμα του εντάγματος σύλληψης για τρομοκράτη για το τρομοκράτη που από την Ιταλία πήγε στον Ηνωμένο Βασίλειο σε δέκα ημέρες αντί χρόνια. Είναι χρησιμότατο πιστεύω το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Αυτό μα το έδειξε αυτό το παράδειγμα. Σε επίπεδο διακυβέρνηση, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση ατόμων κυρίω, μια ελευθερία με την οποία μεγάλωσα, τη θεωρούσα σαν αυτονόητη και θα, ήμουν, θα αισθανόμουν άσχημα αν την έχανα. Λοιπόν, η εδαφική δέσμευση των συστημάτων απόδοση δικαιοσύνη είναι μια πρόκληση και σωστά τίθεται το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξεφύγουμε από αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορούμε να κάνουμε πολλά για να βελτιώσουμε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Διπλή υποχρεωτική υπεράσπιση. Ταυτόχρονη ακροματική διαδικασία όσον αφορά την υπόθεση θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό όπως και απόφαση παράδοσης. Και έχουμε το εργαλείο να κάνουμε αυτό. Αν θέλετε, αν σας αρέσει αμοιβαία αναγνώριση, εγώ δεν λέω ότι μου αρέσει απαραίτητα, αν σας αρέσει αμοιβαία αναγνώριση, είναι μια αρχή η οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Είναι σημαντικό να μην έχουμε αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων που περιορίζουν την ελευθερία και μόνο, αλλά και αποφάσεων που αυξάνουν την ελευθερία. Και απόφαση, ε, η απόφαση πλαίσιο ευρωπαϊκή για την εποπτεία το επιτρέπει αυτό. Η Ευρώπη που είναι θεσμός που έχει ειρηνικό χαρακτήρα και θέλει να αυξάνει την ελευθερία. Λοιπόν, πώς να, εφαρμόζει ένα πλαίσιο που περιορίζει τα δικαιώματα των πολιτών και σε έτσι σε ευάλωτη κατάσταση και δεν έχουμε ανάλογη απόφαση πλαίσιο που να προωθούν κόμματα τα δικά στο Κοινοβούλιο που να εξασφαλίζει την προώθηση και να μην αναγνώριση αποφάσεων που αυξάνουν τις ελευθερίες. Γιατί αναγνωρίζουμε το ένταλμα σύλληψης του εισαγγελέα πιο εύκολα από την απόφαση δικαστού που θα πρέπει να πηγαίνει στο δικαστήριο και να αναφέρεται και να παραδώσει το, το διαβατήριό του μέχρι ότου να είναι έτοιμο το δικαστήριο να εκδικάσει την... απόφαση. Και εκεί θα περιορίζεται για λίγες μέρες. Ενώ τώρα όσο έχει κατάσταση μπορεί κάποιος ύποπτος ε, να κρατείται επί χρόνια σε... Ε, πριν δικαστεί. Λοιπόν, νομίζω τα κάτι μέλη φταίνε περισσότερο δεν εφαρμόζουν σωστά και με τον ίδιο τρόπο τις αποφάσεις πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί στις Βρυξέλλες. Και είναι πολύ κρίμα που το Ευρωπαϊκό Τμήμα Σύλληψη πέρασε το 2002, αλλά το ένταλμα για την εποπτή και τον έλεγχο μόλις το 2009. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες τώρα. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη ε, ε, δεν εξυπηρέτησαν τους πολίτες τους. Διαποφάσισαν ότι οι προτερότητες όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη είναι το σπαθί αλλά επίσης η δικαιοσύνη κρατά από την άλλη και ε, στα σύμβολα που ξέρω και μια μεγάλη ασπίδα για να υπασπίσει τα δικαιώματα. Λοιπόν, το θέμα της επικουρικότητας που αναφέρατε κυρία Μακιντάερ, προσπάθησα στη σύντομη παρουσίαση να τονίσω τον ευρωπαϊκό ρόλο. Βέβαια, η συνεργασία με τα κράτη-μέλη είναι ζωτική σημασία. Ο Ευρωπαίος εισαγγελέα είναι ενδιαφέρον θέμα προς συζήτηση. Μπορούμε να συζητήσουμε την επανάσταση και αυτό τον ενδεχομένως ε, ομοσπονδιακού τύπου ε, φορέα. Σαν Βρετανίδα επίκος δεν έπρεπε να χρησιμοποιώ τη λέξη ομοσπονδιακός. Αλλά καμία ευρωπαϊκή υπηρεσία, όσο και καλούς πόρους έχει, δεν μπορεί να κινείται ανεξάρτητα από τι αρχέ των κρατών μελών. Χρειάζεται πληροφορίε από τα κράτη-μέλη, χρειάζεται συνεργασία με τα κρατη και συνήθω χρειάζεται δραστηριότητα επιτόπου. Λοιπόν, όπω και οι Ιταλικές δομές κατά πολέμηση τη μαφίας βλέπουμε ότι η κεντρική υπηρεσία είναι αποτελεσματική και λειτουργεί μόνο αν έχει υποστήριξη από όλες τις άλλες συνιστώσεις. Είναι ζωτική σημασία να αναγνωρίσουμε ότι ασδήποτε φορές Ευρωπαϊκής Ενώσεως ανεξάρτητα από τις εξουσίες του πρέπει να είναι το κέντρο ενός ιστού και ο ιστός θα καλύπτει και τις αρχές των κρατών μελών και πρέπει να υπάρχουν καλές σχέσεις όσον αφορά τα διάφορα νευραλικά σημεία. Διαφορετικά, οσδήποτε χώρο για το ποινικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα πώ θα συλληφθεί και πώ θα εφαρμοστεί και τι πώ θα έχει, θα λειτουργεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που θέσατε το άλλο θέμα, που είναι κεντρική σημασία, τη κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα τη ποινική δικαιοσύνη. Παρόλο που είμαι νομικό και διδάσκω ε, νομικό δίκαιο, είμαι ε, και ποινικολόγο και ξέρω ότι και η νοτροπία είναι πάρα πολύ σημαντική. Όσο και νομοθεσία. Και βασικό στοιχείο όσον αφορά την άπτυξη σχέσεως μεταξύ επίπεδου κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτου σχετίζεται με διαφορετική επίγνωση, νοοτροπία όσον αφορά τους επαγγελματίες του ποινικού δικαίου όταν αντιμετωπίζουν του πολίτες. Τόσο όσον αφορά την, την αρχή της αναλογικότητας του Ευρωπαϊκού Ένταλμα Σύλληψης, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι οι εισαγγελείς παίρνουν διαφορετικές αποφάσεις όσον αφορά την αναλογικότητα έναντι των δικών τους πολιτών, των ημεδαπών και των άλλων, των αλλοδαπών. Νομίζω ότι είναι σφαλμένο αυτό, τη βάση του, όταν εισαγγελέα ασχολείται με ένα ευρωπαϊκό μέτρο, εκείνος ή εκείνοι πρέπει να θεωρούν ότι είναι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ή Ευρωπαίοι αστυνομικοί. Ανεξάρτητα από την υπηκότητα του πολίτου που έχουν μπροστά τους, υπέχουν καθήκον να φροντίσουν τον πολίτη ως Ευρωπαίο πολίτη. Διότι σε αυτή την περίπτωση ένας Γερμανός, Γάλλος, Βέλγος, Βρετανός αστυνομικός ή εισαγγελέα δρά υπό ευρωπαϊκή εντολή, με ευρωπαϊκή δικαιοδοσία. Και έτσι, οσδήποτε φορέας αρμόδιος, δικαστικός ή άλλος, που έχει ευρωπαϊκό κύρος και ιδιότητες, έχει και αντίστοιχο καθήκον ευρωπαϊκό να προστατεύει ονδήποτε ευρωπαίο πολίτη έχει απέναντί του. Χρειάζεται αλλαγή συνειδητοποίησης, συνείδησης που μπορεί να επιτευχθεί με κατάρτισης. Λοιπόν, Γάλλο. Ε, λοιπόν, υπάρχει το γαλλικό, γερμανικό, ισπανικό σύνταγμα που, που, στο οποίο υπακούν οι διάφοροι εθνικοί εισαγγελεί, αλλά όταν έχουν και κάποια ευρωπαϊκή θέση και καθήκον, έχουν ευρωπαϊκό καθήκον, πρέπει να αντιμετωπίζουν καταλήλα και του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστώ πολύ. Και... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δόκτωρ Βέιτ και Δόκτωρ Μπάουμαν. Ε, ενημερώνω του συναδέλφου ότι έχουν το φυλάδιο αυτό, το έντυπο αυτό για την ποινική δικαιοσύνη και είναι το καλύτερο από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Σας ευχαριστούμε. Ήταν πηγή έμπνευση στα λόγια σας μέχρι τώρα. Σταματούμε εδώ. Προβλέπετε ψηφοφορία για τις 11.45 και ως συνήθως βλέπω να μπαίνουν συνάδελφοι για την ψηφοφορία μαζικά. Στα διακόπτω λοιπόν για τρία λεπτά. 11.45 και αρχίζουμε τις ψηφοφορίες και παρακαλώ να μην αποχωρήσει κανείς, απλώς να κάνετε χώρο για αυτούς που θέλουν να μπουν. Και ετοιμαστείτε. Ετοιμάστε και τις ηλεκτρονικές σας κάρτες παρακαλώ. Βλέπω ότι μερικοί από σας τρέξατε να φέρετε την κάρτα σας και γι' αυτό άφησα ακόμα ένα περιθώριο για να ξεκινήσουμε. Πιστεύω τώρα να είστε έτοιμοι όλοι. Πάρτε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες και ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Δεν είναι περίπλοκες, αλλά είναι πολλές. Και πρέπει να συγκεντρωθούμε. Στο σημείο 17 λοιπόν. Έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη εξ νόμου Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και των κρατών μελών τη, αφενό, και των δημοκρατιών τη Κώστα Ρίκα, του Ελσαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, τη Ονδούρα, τη Νικαράγουα και του Παναμά αφετέρου, όσον αφορά το άρθρο 49, παράγραφο 3. Η κυρία Ρενάτε Βέμπερ δεν είναι παρούσα εισηγήτρια. Συνεχίζουμε όμω με την ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ψηφοφορία του κειμένου. Όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει ηλεκτρονικά παρακαλώ η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Τι αποτέλεσμα. 40 υπέρ. 5 κατά. Ουδεμία. Αποχή. Ορίστε. Έχετε ξεχάσει την κάρτα σας, έχετε πρόβλημα με την κάρτα. Χωρίς μικρόφωνο η απάντηση δυστυχώς δεν έχω. Σας σημειώνουμε πάντως. Υπέρ, υπέρ, α, υπέρ, υπέρ, καλά. 41 ψηφί υπέρ, 5 κατά, ουδεμία αποχή και εγκρίνεται ως εκ τούτου. Περνώ στο επόμενο θέμα. Την πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τι τρίτε χώρε, η υπηκόη των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση και τη για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και τρίτε χώρε, οι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, χωρί τροπολογίε, όπω έχει το κείμενο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν αρχίζει. Η πρώτη ήταν της Μολδαβίας. Λοιπόν, πέρασε η συνεδρία της ψηφοφορίας και 45 υπέρ 2 κατά. Μία αποχή εγκρίνεται κυρία Φαζόν. Η εντολή τώρα για την έναρξη των διαπραγματεύσεων αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Plus. 46 υπέρ, 2 κατά, ούτε μία αποχή εγκρίνεται. Και πάμε πάλι στο ίδιο θέμα. Όχι, όχι, όχι, το είδα, το είδα, το είδα. Το είδα. Σημείο 19. Έλεγχος των προσώπων στο εξωτερικά σύνορα βασιζόμενο στη μονομερή αναγνώριση από την Κροατία και την Κύπρο ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις για το σκοπό της διέλευσης από την επικράτειά τους ή όταν υπάρχει πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών με την κυρία Τάνια Φαγιόν και πάλι δεν είναι εδώ καλώς, άρα δεν θα λάβει και το λόγο και ψηφίζουμε το κείμενο του τριμερούς διαλόγου. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Τι έγινε. Εντάξει, έκλεισε η ψηφοφορία 47 υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Ομόφωνα λοιπόν. Το επόμενο θέμα. Συμφωνία πλαίσιο εταιρική σχέσης συνολική συμφωνία πλαίσιο εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και των κρατών μελών τη Αφενό και τη Δημοκρατία τη Ινδονησία Ευετέρου όσον αφορά συζητήματα που αφορούν την επανεισδοχή. Έχουμε την κυρία Άννα Γκόμε, συγγήτρια. Ψηφίζουμε το κείμενο. Αρχίζει η ψηφοφορία χωρί τροπολογίε. Το σχέδιο εκθέσεω. Πέρα τη ψηφοφορία. 43 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά, μία αποχή και εγκρίνεται. Προχωρώ Point number 21, are you sure? Σημείο 21, αυτό είναι λέτε, στο 21 είμαστε. Έχουμε εδώ, Μαρία Γκαμπριέλ. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 21. Απαλλαγή 2012. Γενικός προϋπολογισμός. Κυρία Ρόιτο. Δεν θέλετε να λάβετε το λόγο. Αρχίσουμε την ψηφοφορία. Point number 21. I mean, I... Ψηφίζουμε το σημείο 21. Και εγώ τα έχω μπερδέψει λίγο, γιατί έχω ένα κατάλογο ψηφοφοριών με έναν αριθμό τροπολογιών κτλ. Εσείς τι έχετε, κατάλογο ψηφοφοριών, ποια είναι η κατάσταση. me just a second. There seems to be... Με συγχωρείτε ένα λεπτάκι, γιατί βλέπω να υπάρχει μια σύγχυση προς το κατάλογο των ψηφοφοριών. Ακόμα και εγώ έχω μπερδευτεί με διορθώνει γραμματεία και μου λέει ότι πάμε στο 21. Αλλά εμένα δεν μου το λέει αυτό ο καταλόγος του ψηφοφοριών. Εσείς τι έχετε. Ναι, ναι. 21 απαλλαγή έχετε εσείς. Εμείς όχι. Απαλλαγή ψηφίζουμε τώρα. Listen, just, just a second. I'm, trying to, trying to have it myself. Καλά, να το βρω τότε κι εγώ. Αφού πάμε στην απαλλαγή. I see, I see. Α, μάλιστα, το βρήκα. Το βρήκα, το βρήκα. Είναι τη σελίδα. Καλώ, το βρήκα. Ρόιτοβα. Απαλλαγή γενικού προπολογισμού. Αρχίζουμε και την ψηφοφορία χωρίς τροπολογίες. Πέρασε. 48 υπέρ μία αποχή. Καμία ψήφος κατά εγκρίνεται. Απαλλαγή για την εκτέλεση του προπολογισμού της ε, υπηρεσία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ψηφίζουμε χωρίς τροπολογίες. Πέρασε. 47 υπέρ καμία ψήφος κατά, δύο αποχές. Απαλλαγή τώρα για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 2012 με την κυρία Ρότεβα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Closed. 47. Πέρασε. 47 υπέρ, μία κατά, μία αποχή. Συνεχίζω με τις υπηρεσίες, οργανισμούς, τέλος του προπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό του 2012, επιδόση δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος, με την κυρία Βερονίκ Ματιέ Ουλιόν. Μία τροπολογία υπάρχει, η υπαριθμών 1, ας την ψηφίσουμε παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη όπως τροποποιήθηκε το κείμενο, το αρχικό κείμενο, ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρας. 46 υπέρ, μία κατά, δύο αποχές. Κυρία Βερονίκ Ματσιού, και πάλι απαλλαγή για τον προπολογισμό της Eurojust και δεν έχουμε τροπολογίες, ψηφίζουμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Σαραντεπτά υπέρ. Μία κατά. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Απαλλαγή. Χωρίς τροπολογίες. Αρχίζουμε. Πέρας. 48 υπέρ. Ομόφωνα λοιπόν και προχωρώ στην απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Europol με την κυρία Βερονίκ Ματσιου Ιού. Τροπολογίες υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο. Αρχής προφορία. Πέρασε. 48 υπέρ. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Και περνώ την ε, υπηρεσία Frontex για την ε, συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα με δύο τροπολογίες. Πρώτη υπαριθμόν 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Αρχίζει η ψηφοφορία ονομαστικά. Πέρασε. 48. Μία ψηφο κατά, καμία αποχή και εγκρίνεται. Έχουμε ακόμα ένα-δύο θέματα. Απαλλαγή. Απαλλαγή ε, Ακαδημίας Αστυνομίας. Η ΣΥΠΟΛ. Κυρία Βερονίκ Ματιέ. Βλέπω κάποιες ε, γλωσσικού χαρακτήρα τροπολογίες, αλλά υπάρχει μια τροπολογία της Ιδρίας η υπαριθμόν 3. Όχι. Ψηφίζουμε υπέρ της τροπολογίας Αυτό σας είπα. Αυτό ή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το συνολικό κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρασε. 43 υπέρ 5 κατά μία εποχή. Εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία. Το Γραφείο Υποστήριξη του Ασύλου. Η συγγήτρια κυρία Ματιό, δεν υπάρχουν τροπολογίε. ψηφίζουμε το κείμενο, συνολικά ψήφο. ηλεκτρονική άρχεται. Πέρασε. 47 υπέρ, μία ψήφο 48 μάλιστα, μία κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. Και τώρα... Το σημείο 31. Κατάλογος τρίτων χωρών, των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να έχουν ε, βίζες όταν διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί οι οποίοι εξαιρούνται από αυτόν τον κανονισμό. Κύριε Γκάμπριελ, θέλετε να λάβετε το λόγο. Όχι, δεν θέλετε. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώ θέλω να πω στου συναδέλφου. τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν πρωτοφανή συμφωνία να συνάψουμε. Μετά από τριμερή διάλογο πετύχαμε συμφωνία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συμβουλίου και η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας ε, ήδη είχε τοποθεθεί από αυτού τον Νοέμβριο. Να επενθυμίσω τα βασικά σημεία. Έχουμε 16 χώρες ΑΚΕ που θα εξαιρούνται από τη θεώρηση. Έχουμε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έχουμε το Περού και την Κολομβία που θα μεταφερθούν στο θετικό κατάλογο μετά από μια αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό αντιστοιχεί απόλυτα σε αυτά που ψηφίσαμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή των συναδέλφων επί άλλου σημείου που για μας είναι κρισίμου σημασία για τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή τα κριτήρια που τώρα και στο εξή θα εμφανίζονται όχι σε τελογικές σκέψεις αλλά σε άρθρο, πρώτο άρθρο, πάντα η αξιολόγηση θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά περίπτωση, αλλά τώρα πλέον θα υπάρχουν τρία κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη. Το, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο τουρισμό και το εξωτερικό εμπόριο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα θέση του Κοινοβουλίου που πάντα ε, την υπερασπιστήκα και εγώ και οι ηγητέ και τους ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ο τουρισμό και το εξωτερικό εμπόριο προστήθηκαν σαν κριτήρια από το Συμβούλιο. Τέλο, τελικό σημείο, το δικαίωμα ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βούληση αυτή εξ αρχή να έχει τακτικό διάλογο μαζί μα μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει κάποια δήλωση που θα επιβεβαιώσει ότι τακτικά θα ενημερωνόμαστε όσον αφορά τις ε, τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επίτροπη, το Συμβούλιο και κυρίως την Ελληνική Προεδρία για όλες τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για ένα θέμα που τελικά ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης διότι μπορέσαμε να υπερασπιστούμε μια θέση ισχυρή του Κοινοβουλίου για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο πρέπει να θυμηθείτε συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία και τέλο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κατρίνη Ιμπέρ τη Γραμματεία Ενώπιον των Συναδέλφων γιατί χωρί τι γνώσει αυτό το θέμα δεν θα μπορούσε να προωθηθεί εντό των προθεσμιών που θέλαμε να τηρήσουμε και που σεβόμαστε τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ για τη δουλειά σα, Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για θεσιμότητά σα και τις εις βάθος εξηγήσεις που δώσατε όσον αφορά την ε, συμφωνία που ψηφίζουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του τριμερού διαλόγου. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα, έτσι. Υπέρ. Έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρα αυτή. 49 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή, οπότε εγκρίνεται και ευχαριστούμε να σας υπενθυμίσω ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα υποβληθούν στην Ολομέλεια. Ψηφοφορία θα γίνει στην πρώτη σύνοδο του Απριλίου. Καλώς, σας ευχαριστώ όλους. Προχωράμε, έχουμε ακόμα μια ψηφοφορία, η οποία είναι και η μεγαλύτερη. Σήμερα στην πρωινή συνεδρίαση έχουμε να ψηφίσουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την επίτευξη συνδεδεμένης υπήρου μέσω τροποποίησης οδηγιών και κανονισμών. Ο κύριος Σαλβαδόρ Σεδόν είναι ο εισηγητής. Δεν έχετε σχόλιο. Καλώς, μπορούμε να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε. Είναι μεγαλύτερη από την πιο μακροσκελή από τι προηγούμενε. Τροπολογίες 45 και 46 είναι ταυτόσιμες. Ποιο είναι κατά, ποιος είναι υπέρ Ποιό είναι υπέρ, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρο, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 47, υπέρ, κατά, απόχε, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. 49, καλός έλεγχος εγώ δεν τα εγκρίνεται, αλλά κάνουμε επαλήθευση, ίσως έχετε δίκιο. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Πέρας. 26 υπέρ, 25 κατά, μικρή διαφορά. Πολύ μικρή διαφορά, αλλά εγκρίνεται. 49 λοιπόν και 50 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 51 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι το ίδιο ισχύει όπως και με την προηγούμενη αν θέλετε να κάνουμε επαλήθευση τον ίδιο συσχετισμό είδα την ίδια πλειοψηφία υπέρ γίνει έλεγχος λοιπόν τώρα για την 51 έρχεται η ψηφοφορία Closed. Πέρας ψηφοφορίας. Αυτή τη φορά είναι αντίθετο το αποτέλεσμα. Έκανε λάθος κάποιος. 25 υπέρ 26 κατά απορρίπτεται. Εντάξει. 52, 53, 54, 55 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές δεχτεί. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 58 άρχεται η ψηφοφορία το ΕΛΚ έχει ένα που ψηφίζει παραπάνω. Πέρασε. 26-25 εγκρίνεται. Οκτώ και 59 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές 60, 61 και 62. Υπέρ. Κατά. Από χέρια συγκρίνονται. 63. Εκπίπτει 63. Ούτε η 9 πρέπει να ψηφιστεί. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 66. Άρχεται η ψηφοφορία. περασε με 29 απόρριπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβαστη 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 77. Άρχεται η ψηφοφορία για την 77. Πέρασε. 19-29 απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίτη. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απεσύρθη 11, 88, 89 και 90 ταυτόσιμες. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεν γίνονται δεκτές. 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 98, 99 και 100 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Έλεγχος για τις 98, 99 και 100. Πέρας προφορία. 25 υπέρ 26 κατά απορρίπτονται. Συνδέονται κάπως αυτές οι τροπολογίες μεταξύ τους. Πάμε στην τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Η 12 ανεκρίθη, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Ας ελέγξουμε. Τροπολογία 12. Υπε, ε, ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται, απορρίπτεται, ναι. Τροπολογία 23, 13, υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 101, 102 και 103 που είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές έλεγχος 118 έρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας 25-26 απορρίπτεται 122 και 123 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 129 υπέρ κατά αποχές δεχτεί 130 υπέρ 129 έλεγχος έλεγχος ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται πράγματι 130 130 υπέρ κατά αποχές το ίδιο αποτέλεσμα εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για την 131 άρχεται πέρας 25-26 απορρίπτεται Υπάρχει κάποιος ο οποίος αλλάζει συνέχεια γνώμη, λέει ο πρόεδρος. Και τροποποιεί τις πλειοψηφίες. Απερίφθη λοιπόν. 132 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Έλεγχος για την 132, ναι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 25-26. 133. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο. Έλεγχος. 133. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. ως 5.26 εγκρίνεται. Εtiολογικές σκέψεις και αναφορές. Έχουν αποσυρθεί οι ορισμένε τροπολογίε. 22 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 23. 23 έλεγχος. πέρασε. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 30 έλεγχος για την 4 ειτε ελεγχο έλεγχος άρχεται πέρας 33-18 εγκρίνεται η 30 εκπίπτει ω αποτέλεσμα Εκπίπτει, ναι, ναι, πράγματι. Οι 30 και 29 εκπίπτουν. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για την 31. Πέρας ψηφοφορίας. με ισοψηφία απορρίπτεται. Αυτός που μετακινείται κράτησε στάση εποχής. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά, αποχές δεκτή. 33, υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Το σύνολο του κειμένου τώρα, όπως έχει τροποποιηθεί. Κύριε Τάνοκα, χωρίς μικρόφωνο η ομιλητή. Μπορείτε, μπορούμε να ψηφίσουμε την τροπολογία 31. 31. It doesn't, I your vote η ψήφος σας δεν θα αλλάξει. Θα μπορούσε. Μία ψήφος θα μπορούσε να το αλλάξει. Ναι, δεν το βλέπω λέει ο Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει βάση του εσωτερικού κανονισμού. Λυπάμαι, δεν προβλέπετε. Διεξήχθη η ψηφοφορία, λυπούμε γι' αυτό. Τελείωσε, βγήκε αποτέλεσμα. Τελική ψηφοφορία του αποποιημένου κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. 48. Μηδέν αποχές, μηδέν αντιρρήσεις, ομοφωνία, συγχαρητήρια λοιπόν συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ όλους, σταματάμε για την ώρα, στις 3 συνεχίζουμε. Α, ζητώ συγγνώμη, η κάρτα μου δεν μπήκε στο μηχάνημα στην τελευταία ψηφοφορία. Μπορείτε να λάβετε υπόψη την ψήφο μου. Θα προσθέσουμε ένα συν, μια θετική ψήφο. Λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Στις 3 τα ξαναλέμε. Καλή όρεξη. Γεια σας.